Είναι επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι και καλεσμένοι. Μια και απουσιάζει ο κύριος Κλίντς, θα έχω εγώ την τιμή να προεδρεύσω στο σημερινό εργαστήριο για την επίπτωση της κρίσης στα νέα κράτη-μέλη. Χαίρομαι για τη διοργάνωση αυτού του ειδικού σεμιναρίου που αφιερώνεται σε αυτό το θέμα, γιατί οι οικονομίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι αυτές που χτυπήθηκαν πιο στιγνά από την κρίση. Και ταυτόχρονα πολλές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις στρατηγικές πάταξεις της κρίσης και τα μέτρα ανάκαμψης ε, επικεντρώνονται γύρω από τις ε, χώρες της ζώνης ευρώ, ενώ οι νεοεισερχόμενες στην Ένωση χώρες είναι αυτές που είναι πιο ευάλωτες στην κρίση. Παρόλο που Μερικές από τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη είχαν από τι πιο αυστηρέ και υγιεί δημοσιονομικέ πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα στην Ολομέλεια προκειμένου να αναζωογονήσουμε τις οικονομίες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπη και ω εκλεγή βουλευτή από νέα χώρα Χαίρομαι για την αλληλεγγύη που εκφράστηκε προς τις νέε χώρε μέλη και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την κατανόησή τους ω προς το βαθύτατο αντίκτυπο που έχει κρίσει στις οικονομίες μας και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τη στην αηφόρο ανάπτυξη στι νέε χώρε. Βέβαια, όταν υπάρχει θέμα αλληλεγγύη, άσχετα από το αν αφορά ένα νέο ή ένα παλιό μέλος της Ένωσης, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι κάθε χώρα οφείλει να υπομειστεί τις ευθύνες της και να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις τηρώντας ε, τα κοινά κριτήρια για την Ομισματική ένωση. Σήμερα η Επιτροπή μας θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τις ομιλίες και παρουσιάσεις πολλών ε, διακεκριμένων καλεσμένων. Θα έχουμε δύο πάνελ και κάθε καλεσμένος μας θα έχει ένα δεκάλεπτο για να μας παρουσιάσει τις ιδέες του. Κατόπιν θα γίνει συζήτηση. Το πρώτο πάνελ αφιερώνεται στο μακροοικονομικό αντίκτυπο, την παρακολούθηση και εποπτεία των ε, μακροοικονομικών πολιτικών. Ο κύριος Στανίσλαφ Κομούκα, ο τρίτος καλεσμένος, έχει κολλήσει στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Μπλοκαρίστηκε εκεί και δυστυχώς δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στο σεμινάριο, αλλά μας έστειλε ένα πεντασέλιδο έγγραφο και είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει γραπτός στις ερωτήσεις που μπορείτε να του στείλετε επί της παρουσίασής του. Ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο Φίλιπ Κιρέμαν που είναι προϊσταμένος της μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΦΗΝ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο της ε, Μονάδας Παρακολούθησης των Εθνικών ε, Δημοσιονομικών Εξελίξεων στην εξωτερική ε, χρηματοδότηση. Η δεύτερη ευρύτερη είναι η κυρία Καταρζίνα Σμίτκοβα, εκτελεστική διευθύντρια του Τμήματος Οικονομικής Έρευνας και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας και ο κύριος Ζολ Ντάρβας από, ε, την ε, Bridge Research Fellow. Φυσικά και οι, δύο καλεσμένοι μας, οι τρεις καλεσμένοι μας θα δώσουν γραπτό στις ομιλίες τους. Στο δεύτερο πάνελ θα εξετάσουμε το ρόλο της ε, στρατηγικής συνοχής. Και θα ακούσουμε δύο μιλητές, τον κύριο Πίτερ Χάιλ και τον Φάμπιαν Ζουλέγκ. Στο πρώτο πάνελ θα εξετάσουμε τις αιτίες και τις επιπτώσεις της κρίσης στις νέες χώρες μέλη, καθώς ε, και τις απόψεις των εισηγητών μας για την ε, συνεργασία ως προς την παραγωγή εντός και εκτός Ευρωζώνης και τη δυνατότητα διεύρυνσης της Ευρωζώνης. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Φίλιπ Κέρεμανς, που θα μας παρουσιάσει τις δικές σου απόψεις για τον αντίκτυπο της κρίσης στα νέα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σας. Και θα ήθελα κάποιος να βοηθήσει με το PowerPoint.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 χωρίσει την ομιλία μου σε πέντε θέματα με τα βασικά μου μηνύματα. Όπως βλέπετε δεν πρόκειται για μια διεξοδική παρουσίαση της κρίσης, για το περί τίνος πρόκειται και ποια είναι η επίπτωση της κρίσης σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα επικεντρωθώ σε ορισμένα πιο συγκεκριμένα θέματα. Το πρώτο θέμα αυτό το είναι που ανέφερε και η Πρόεδρος, δηλαδή η επίπτωση της κρίσης στα νέα κρατημέλη που ήταν ισχυρότερη από ό,τι στα παλιά κρατημέλη. Και εκεί θα εστιαστώ σε μία απάντηση πολιτικής που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η βοήθεια σε θέματα ισολογισμού πληρωμών, ισοζυγίου πληρωμών στα νέα κράτη-μέλη. Αυτή, κατά τη γνώμη, ήταν μια επιτυχής απάντηση πληρωμων στα νεα κρατη αυτη κατα τη Επίσης, οι ε, τράπεζες έπαιξαν, σημαντικό ρόλο στα νέα κράτη-μέλη. Συνέβαλαν στην ε, ανάπτυξη, στην οικονομική εφορία αλλά και στην, ε, ε, στην κρίση που ακολούθησε. Γι' αυτό και θεσπίστηκε η πρωτοβουλία, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για, την για το τραπεζικό συντονισμό προκειμένου οι ξένες τράπεζες που εγκαταστάθηκαν στη χώρα αυτή να παραμείνουν τα χρήματα που δόθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα αυτή να μην ε, διαρρεύσουν. Τέταρτο θέμα. Ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απέναντι στις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ. Και επίσης ποιοι είναι οι μηχανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες εντός της Ευρωζώνης σε σχέση με τους μηχανισμούς για τις χώρες εκτός της Ευρωζώνης και το πέμπτο θέμα είναι τα συμπεράσματα και οι μελλοντικέ προκλήσεις ή οι προκλήσεις που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Τα περισσότερα νέα κράτη-μέλη ε, βίωσαν μία ισχυρότερη ύφεση από ό,τι οι παλιές χώρες, κυρίως στα χρηματοπιστωτικά και εμπορικά θέματα. Ο αντίκτυπος γενικώ ήρθε κάπως αργότερα, σε σχέση με τις παλιές χώρες μέλη, αν και στις βαλτικές χώρες συγκεκριμένα η κρίση ε, έγινε αισθητή ήδη από τα πρώτα στάδια της. Χαρακτηριστικό της επίπτωσης της κρίσης στις νέες χώρες μέλη είναι ότι η αίσθηση του κινδύνου έγινε μεγαλύτερη, οξύτερη στις νέες χώρες μέλη. Και ένας από τους λόγους ε, το ότι ένιωσαν αυτό το σοκ περισσότερο στις νέες χώρες ε, μέλη είναι ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν σε επίπεδο πολιτικών προς τις χώρες αυτές ήταν μάλλον περιορισμένες εμβέλειες. Επίσης, ένα άλλο ειδικό χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική διόρθωση των τιμών ακινήτων στις νέες χώρες. Η παρακμή της οικονομικής δραστηριότητας ε, στην Ευρωζώνη ήταν πιο ήπια και είχε, ήταν πιο εξαπλωμένη. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία αυτού που σας παρουσίασα προηγουμένως. Δηλαδή, την ε, μείωση στα κράτη-μέλη, την ύφεση από πολύ ψηλά ε, επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης σε πολύ χαμηλά, πρώτα στις νέες χώρες και μετά στην Ευρωζώνη και μία βαθύτερη ύφεση κυρίως στις νέες χώρες μέλη. Ποιες χώρες από τις νέες χώρες μέλη χτυπήθηκαν περισσότερο. Ήταν αυτές που είχαν τις μεγαλύτερες ανισορροπίες εξωτερικές τους ε, χρηματοπιστωτικές ροές, γιατί ήταν περισσότερο εξαρτημένες από εισαγωγές κεφαλαίων για να ενισχύσουν ε, την διόγκωση των πιστοληπτικών αναγκών τους και για λόγους εμπιστευτικότητας, ε, απορρίτου, γιατί τα επίπεδα χρέους που συσσωρεύτηκαν ε, πολύ γρήγορα στις νέες χώρες, επίσης ε, μειώθηκαν ε, οι ροές κεφαλαίου, αυξήθηκαν τα επιτόκια απότομα και δημιουργήθηκαν κάποια χρηματοπιστωτικά κενά στις νέες χώρες. Και χρειάστηκε η επέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία αναχώρα σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της κρίσης και αν υπολογίσουμε το σωρευτικό αντίκτυπο της κρίσης από την εχμή της ανάπτυξης στο τρίτο ε, τρίμηνο πέρυσι, για το οποίο είχαμε πληροφορίες, διαπιστώνουμε ότι το ΑΕΠ συρρυκνώθηκε περισσότερο στις βαλτικές χώρες, στην ε, Λετωνία ε, συρρυκνώθηκε πάνω από 30%, 20% ε, συγγνώμη, και σε ορισμένες παλιές χώρες μέλη η, η, επίπτωση ήταν η ποιότερη. Πάντως, μόνο η Πολωνία δεν βίωσε πολύ οξία ύφεση. Γενικώ και αν δούμε την τελευταία διετία η Πολωνία κατάφερε να διατηρήσει την τελευταία διετία θετική ανάπτυξη. Βλέπετε ότι στις νέες χώρες η επίπτωση ήταν σημαντικότερη από ότι στις παλιές χώρες, με εξαίρεση την Πολωνία, που η ύφεση ήταν η ποιότερη. Μία σημαντική αντίδραση σε επίπεδο πολιτικής είναι αυτό το θέμα της αρρωγής ε, για το ισοζύγιο πληρωμών. Η αρρωγή αυτή εντοπίστηκε κυρίως στις ε, χώρες εκτός Ευρωζώνης. Και όταν μια χώρα ζητά την ε, αρρωγή αυτή στο πληρωμών, θα πρέπει καταρχήν να υποβάλει σχετικό αίτημα και τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία αν θα εγκρίνει αυτό το αίτημα και κατόπιν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται τις λεπτομέρειες και τους όρους των δανείων. Όλα αυτά σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο ό,τι αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εφαρμογή. Και αυτό γίνεται από, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πραγματοποιούνται και κοινέ αποστολές. Μάλιστα υπάρχει ένα ανώτατο όριο 50 δισεκατομμύριων στα πλαίσια αυτής της αρρωγής, ένα κατόφλι που αυξήθηκε από 12 δισεκατομμύρια πριν από μία διετία στο σημερινό κατόφλι των 50 δις. Μόνο η Ουγγαρία, η Λετωνία και η Ρουμανία μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το μηχανισμό αρρωγής για το ισοζύγιο πληρωμών. Εδώ έχετε μια γενική επισκόπηση των αρχικών ποσών που δόθηκαν στις χώρες αυτές, 20 δις στην Ουγγαρία, δηλαδή 20% περίπου του ΑΕΠ, στη Λετωνία 7 δις, τεράστιο ποσό, γιατί αντιπροσωπεύει το 40% περίπου του ΕΠ, και στη Ρουμανία δόθηκαν 20 δισεκατομμύρια, περίπου δηλαδή λίγο λιγότερο από ό,τι στην Ουγγαρία σε ό,τι αφορά το, ποσοστό του ΕΠ. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου. Συνήθως ε, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο συμβάλλει περισσότερο, με εξαίρεση τη Λετωνιακή ήταν σημαντικότερη συνεισφορά της Ένωσης. Στην περίπτωση της Λετωνίας και πάλι υπήρξε και διμερής υποστήριξη από μεμονωμένες χώρες μέλη. Άλλες ήταν ευρωπαϊκές και άλλες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και η Νορβηγία έδωσε το παρόν και ε, έδειξε τιμότητα να δανείσει τη Λετωνία. Και μάλιστα δύο χώρες για λόγους αλληλεγγύης, αλλά και για να δείξουν ότι μπορούν να διαθέσουν τέτοια κονδύλια βοήθειας είναι η Πολωνία, ήταν η Πολωνία, η Εστονία και η Τσεχία, που και αυτές προθυμοποιήθηκαν να δανείσουν στη Λετωνία. Περνάμε μια διάμεση διαφάνεια και έρχομαι σε ένα σημαντικό σημείο που αφορά το ρόλο των διεθνών τραπεζών ιδιαίτερα στις τρεις χώρες ε, που έλαβαν διεθνή χρηματοοικονομική βοήθεια. Αυτές ε, οι χώρες ήταν σημαντικές για την ε, ισορροή κεφαλαίων που έλαβαν, αλλά και για την συμβολή τους στην ανάπτυξη. Και μετά από αυτές τις αρχές κεφαλαίου ήταν σημαντική η οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε. Εδώ φαίνεται η σπουδαιότητα ορισμένων διεθνών ομίλων στις χώρες αυτές και είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές αυστριακές τράπεζες ενεργοποιήθηκαν στην περιοχή και μάλιστα όχι σε μία μόνο χώρα αλλά σε περισσότερες, αλλά και ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε αντίθεση με τις σκανδιναβικές τράπεζες, που ίσως και για γεωγραφικούς λόγους βρίσκονται μόνο στην Λετωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Συντονισμού, περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται κυρίως για ένα διάλογο με τις ε, τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προκειμένου να, υπερ... υπερκεραστεί ένα πρόβλημα συλλογική δράσης που θα οδηγούσε σε μία ε, σε μία φυγή προς την έξοδο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συντονισμός, ε, υπάρχει πρόβλημα στη στρατηγική. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλες οι τράπεζες έχουν συμφέρον, αν βλέπουν την κρίση να πλησιάζει, να σπεύσουν προς την έξοδο, να επαναπατρίσουν τις επενδύσεις και τα κέρδη τους πριν εμφανιστεί η κρίση. Και τι σημαίνει η κρίση, σημαίνει υποτίμηση του νομίσματος, και φυσικά οι τράπεζες έχουν συμφέρον να επαναπατρίσουν τι επενδύσει και τα κέρδη του πριν λάβει χώρα αυτή η υποτίμηση. Γιατί οι τράπεζε ενδιαφέρονται για τη μεγιστοποίηση των κερδών του. Τώρα, για το σύνολο τη κοινότητα, του διεθνεί δωρητέ, την ίδια τη χώρα, αλλά και για όλε τι τράπεζε, για τον τραπεζικό κλάδο, υπάρχει συμφέρον να παραμείνουν δραστήριε στη χώρα, γιατί έτσι θα αποτρέψουν τον κίνδυνο Γι' αυτό και στόχος είναι να ενημερωθούν οι τράπεζες για το κίνδυνο αυτό, να μην δημιουργηθεί ένα αποτέλεσμα ντόμινο και να πιστούν να παραμείνουν στην χώρα με το επιχείρημα ότι θα δρέψουν κέρδη, παρόλο που υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή, αλλά ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, υπάρχει δυνατότητα ε, συμφωνίας και είναι πολύ πιθανό να υπερκεραστεί αυτή η χαλεπή περίοδο στη χώρα αυτή, οπότε θα ακολουθήσει περίοδος ανάπτυξης και διόγκωση των κερδών των τραπεζών. Πρόκειται για μια συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες, γιατί οι κεφαλαϊκοί έλεγχοι δεν μπορούν να επιβληθούν άνωθεν. Βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ισχύουν οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες και μία από αυτές είναι φυσικά και η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Και η εισαγωγή κεφαλαϊκών ελέγχων θα ήταν ένα πολύ κακό μήνυμα και ίσως και αντιπαραγωγικό. Όπως φάνηκε και στον προηγούμενο πίνακα, ήρθαμε σε συνομιλίες με μερικές μονοβασικές τράπεζες και με το διάλογο προσπαθήσαμε να τις πείσουμε. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε με όλες τις επιχειρήσεις ή τους καταναλωτές, γιατί αυτοί είναι πολύ ανομοιογενής και τεράστια ομάδα και δεν νοείται συντονισμός με τέτοια πολυπληθή ομάδα. Και μάλιστα ο συντονισμός αυτός υλοποιείται μέσω μια σειράς συναντήσεων που έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες, στη Στοκχόλμη αλλά και στη Βιέννη. Α, τελείωσε ο χρόνος μου. Εξαντλήθηκε ο χρόνος μου και άρα πρέπει να φτάσω στα συμπεράσματα. Στις συνομιλίες πάντως αυτές, στις συναντήσεις αυτές, προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ε, να παραμείνουν αυτέ οι, χώρες, οι τράπεζες της χώρα, και αν υπάρξει κίνδυνος ε, κεφαλαιοποίησης, ανακεφαλαιοποίησης, να υπάρχει δυνατότητα κάτι τέτοιο. Γίνονται συναντήσεις και στις, ε, με τη χώρα, αλλά και με όλες τις τράπεζες. Τελευταία συνεδρίαση έγινε την περασμένη Παρασκευή για τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σερβία που δεν είναι φυσικά ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί κονδύλια, δάνεια. Εμπίπτουν δηλαδή σε αυτή την πρωτοβουλία του συντονισμού. Και η επόμενη σημαντική συνεδρία θα γίνει στην Αθήνα στα μέσα Μαρτίου. Αυτή είναι η εξέλιξη για την ε, έκθεση στον κίνδυνο. Πάντως με την πρωτοβουλία συντονισμού αλλά και με την απλή παρουσία των τραπεζών αυτών στις νέες χώρες μέλη κατάφεραν οι χώρες αυτές να ξεπεράσουν την κρίση γιατί οι νέες τράπεζες, οι ξένες ελλοδαπές τράπεζες φρόντισαν ε, να παραμείνει η έκθεση και να γίνει ανακεφαλαίωση, η ανακεφαλαίωση των θηγατρικών τους και επίσης ε, δεν χρειάστηκαν τόσα κρατικά κονδύλια, τόση κρατική επέμβαση όσο στην Ευρωζώνη. Και φαίνεται από τον πίνακα αυτό ότι στην Ευρωζώνη οι, οι εγγυήσεις, ε, η κρατική παρέμβαση ήταν πολύ πιο σημαντική από ό,τι στις νέες χώρες μέλη. Και αυτό ίσως οφειλόταν στο ότι στις νέες χώρες ε, ε, ήταν πιο αξία η κρίση, αλλά ίσως και επειδή στις ε, νέες χώρες οι αλλοδαπές τράπεζες διαδραμάτισαν καλύτερο το ρόλο τους. Έχω και μερικές διαφάνειες για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μηχανισμό αρρωγής, αλλά δυστυχώς έχω ξεπεράσει την ώρα μου. Οπότε θα υποβληθούν και ερωτήσεις σχετικά, οπότε εκεί μπορούμε να επανέλθουμε στις διαφάνειες. το συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε με θετικό τρόπο, αλλά παραμένουν κάποιες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις που θα σας υποβληθούν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Σμιτροβά, που θα μας παρουσιάσει τις ιδέες της ε, από την σκοπιά της Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στο ενδιαφέρον εργαστήριο. Τρία είναι τα μηνύματα που θα ήθελα να περάσω στην παρουσίασή μου, λίγο διαφορετικά από αυτά του Φίλιπ και θα συζητηθούν στο τέλος. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι και οι νέες χώρες μέλη και οι παλές χώρες μέλη είναι πολύ ανομοιόμορφες ομάδες. Δεύτερο μήνυμα ότι οι χώρες μέλη που επλήγησαν από την κρίση είναι κυρίως χώρες όπου ένα συνδυασμός μακροοικονομικών ε, και χρηματοπιστωτικών σταθεροποιητών υπήρχαν, έγινε συνδυασμός δηλαδή και μειώθηκε έτσι η κρίση. Τρίτο μήνυμα είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις μπροστά μας διότι οι παράγοντες που την προκαλούν, την κρίση, είναι περίπλοκοι και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε εύκολα από αυτούς. Θα πρέπει να του αντιμετωπίσουμε λοιπόν με ένα περίπλοκο ε, μείγμα πολιτικών. Πρώτα λοιπόν για την ετερογένεια της ομάδας των νέων χωρών μελών, η οποία από πρώτη άποψη φαίνεται να επλήγησαν οι νέες χώρες μέλη βαρύτερα από τις παλαιές, γιατί βλέπουμε στην διαφάνεια αυτή περισσότερο κόκκινο χρώμα στις νέες χώρες μέλη και οι κόκκινες αυτές γραμμές δείχνουν τις χώρες εκείνες οι οποίες έχασαν παραπάνω από 5% από το καθάριστο εγχώριο προϊόν το 2009 όμως ορισμένες από τις χώρες αυτές είναι πάρα πολύ μικρές. Και όπως είπε ο Φίλιπ στην ομάδα των νέων χωρών μελών έχουμε και την Πολωνία, η οποία είναι η μοναδική χώρα μέλος η οποία έδειξε θετική εξέλιξη. Αν πάρουμε λοιπόν τους μέσους όρους του πληθυσμού των νέων χωρών μελών και των παλαιών χωρών μελών και επίσης των χωρών της ζώνης ευρώ και αυτών που δεν είναι στην ζώνη ευρώ, θα δούμε ότι ο πληθυσμός των χωρών μελών, επλήγει, όλων αυτών των χωρών μελών, επλήγει περίπου με τον ίδιο τρόπο από την κρίση. Κατά κεφαλήν δηλαδή, τα αποτελέσματα είναι πολύ παρόμοια και στις νέες και στις παλαιές χώρες μέλη. Και αυτό καταδεικνύει ότι είναι πολύ ανομοιογενής η ε, ομάδα των νέων χωρών μελών. Δεν είναι λοιπόν τα ίδια για όλες. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λέμε πώς επλήγησαν οι νέες χώρες μέλη σε σχέση με τις παλαιές. Ο λόγος είναι ότι αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης της ε, κρίσης από τη μια χώρα στην άλλη. και ενισχύουμε και την εντύπωση αυτή και απέναντι στις αγορές ότι όλες ε, οι χώρες αυτές μέλη, νέες χώρες μέλη δηλαδή εμπλήξαν με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να ρίξουμε μια βαθύτερη ματιά για να δούμε ποιες χώρες ή ποιες υποομάδες χωρών έχουν διαφορετική ε, αντιμετώπιση. Ο λόγος της ετερογένειας ε, της ομάδας αυτής, δεν είναι ένας λόγος, είναι πολλοί. Προσπάθησα να τους χωρίσω σε δύο ομάδες. Υπάρχουν ορισμένοι μακροοικονομικοί παράγοντες που είναι διαφορετικοί στις νέες χώρες μέλη σε σύγκριση με τις παλαιές και ορισμένοι παράγοντες της ε, οικονομικής σταθερότητας. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες περιλαμβάνουν για παράδειγμα τους μεγάλους οφιλέτες τις μεγάλες ε, οφειλέτριες χώρες οι οποίες είναι πιο τρωτές από την κρίση. Όμως όλες οι νέες χώρες μέλη δεν είναι μεγάλες οφειλέτες, δεν έχουν μεγάλα χρέη δηλαδή. Και έχουμε και εκείνες οι οποίες έχουν ε, σκληρές, άκαμπτες ισοτιμίες δηλαδή, είναι σε λιγότερο ευνοϊκή θέση από εκείνες οι οποίες έχουν κειμενόμενες ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σε ό,τι αφορά τους μακροοικονομικούς παράγοντες σταθερότητας, θα δούμε ότι σε ορισμένες νέες χώρες μέλη τα νοικοκυριά είναι αποταμιευτές. Έχουν λοιπόν περισσότερες, περισσότερες καταθέσεις και ενισχύουν έτσι τον τραπεζικό τομέα. οι οποίες μπορούν μετά να προσφέρουν δάνεια. Επομένως αυτές οι χώρες δεν εξαρτώνται τόσο πολύ από διαμεθοριακές μεταφορές κεφαλαίων. Φαίνω το παράδειγμα της Σλοβακίας και της Τσεχίας, που και οι δύο αυτές χώρες είναι αποταμιεύτριες κατά, κατά, κατά αυτή την έννοια. Ο δεύτερος παράγοντας οικονομικής σταθερότητας είναι ότι οι εγχώριες οι οικονομικές και νομισματικές πολιτικές είναι συντηρητικέ και σταθερές. Υπάρχει και η διαφάνεια που δείχνει πώς επηρεάζουν οι παράγοντες αυτοί με διαφορετικό τρόπο τις διάφορες χώρες. Θα δείτε δύο εικόνες εδώ σύγκρισης νέων χωρών μελών με άκαμπτες ισοτιμίες σε αντιστοιχεία με αυτές που έχουν ε, κειμενόμενες ισοτιμίες και θα δείτε στην πρώτη ομάδα, η πρώτη υποομάδα καλύτερα, η οποία είχε τάση περισσότερο να κάνει μεγάλα εξωτερικά χρέη και, χρέη και να ξεπεράσει το 60% του ΑΕΠ, ενώ οι άλλες χώρες ήταν λιγότερο ευάλωτες από την οικονομική κρίση. Παρόμοια κατάσταση και στις τιμές της στέγης που δεν ήταν το ίδιο σε όλες τις νέες χώρες μέλη, δεν υπήρξε δηλαδή αυτή η φούσκα των τιμών των χωρών μελών, εκεί όπου ήταν άκαμπτες ισοτιμίες, οι συναγματικές ισοτιμίες, ήταν πιο ε, λιγότερο καλή η κατάσταση των αγορών και για τη στέγη. Εάν εξετάσουμε την ομάδα των παλαιών χωρών μελών βλέπουμε περίπου την ίδια εικόνα. Σε ορισμένες χώρες όπως Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία βλέπουμε τιμές στέγης που αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό και μεγάλο εξωτερικό χρέος, το οποίο επίσης αυξάνεται με, μεγάλο, με ρυθμό. Και γι' αυτό το λέω ότι δεν είναι μόνο οι νέες χώρες μέλη αυτές που επλήγησαν από την κρίση. ό,τι αφορά τους παράγοντες οικονομικής σταθερότητας, ο πιο σημαντικός δείκτης κατά τη γνώμη μου είναι η αναλογία δανείων με καταθέσεις. Θα δείτε τις οριζόντιες γραμμές που δείχνουν το μέσον όρο της Ευρωζώνης είναι ανάμεσα στο 25 και 75% και θα δείτε ορισμένες νέες χώρες μέλη όπως την Τσεχία και την Σλοβακία που είναι αληθινές αποταμιεύτριες, δηλαδή έχουν περισσότερες αποταμιεύσεις από ό,τι χρειάζεται καν, δηλαδή πλεονασματικές, για, τα, ε, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν, μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν δάνεια από τις τράπεζες δηλαδή. Και στη δεξιά πλευρά βλέπετε τις βαλτικές χώρες, οι οποίες δεν κατάφεραν να χρηματοδοτήσουν τα εγχώρια δάνεια από τα, από τα τους, από τις καταθέσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ορισμένε νέε χώρε μέλη οι οποίε βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση γιατί δεν εξαρτώνται από διαμεθοριακές κινήσει κεφαλαίων. Όπω είπα επίση η αξιοπιστία των εσωτερικών, των εχωρίων πολιτικών ήταν σημαντική κατά τη διάρκεια τη κρίση. Βλέπετε στην εικόνα αυτή την έκθεση σε εξωτερικά δάνεια, σε αλλοδαπά δάνεια δηλαδή, θα δείτε για ορισμένε χώρε, όπω την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία ότι η ε, τα νοικοκυριά δεν έχουν δανειστεί σε ξένο νόμισμα καθόλου. Ενώ, για παράδειγμα, άλλες παλιές χώρες μέλη, όπως η Αυστρία, το έχουν πράξει αυτό. Και βέβαια, σε χώρες όπου τα νοικοκυριά προτίμησαν δάνεια σε εγχώριο νόμισμα, δεν εξαρτήθηκαν από αλλοδαπό νόμισμα. Και αυτά είναι δείκτες που μας δείχνουν ότι οι χώρες που δεν το έπραξαν αυτό είναι πιο ευάλωτες, διότι όπως είπα ήταν ε, εκτεθειμένες σε διακυμάνσεις ε, των ε, συναλλαγματικών ισοτιμιών. το τελευταίο, η τελευταία διαφάνεια, η τελευταία εικόνα δείχνει την αναλογία της θέσης των ε, τραπεζών σε σχέση με το ΑΕΠ. Πάλι βλέπετε τις οριζόντιες γραμμές που δείχνουν ορίζουν τον χώρο της Ευρωζώνης. Θα δείτε ότι ορισμένες χώρες είναι συγκρίσιμες σε ό,τι αφορά την έκθεση του τραπεζικού του τομέα σε ε, κινδύνους που προέρχονται από την Αλοδαπή. Ορισμένες χώρες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες, ο τραπεζικό, η τραπεζική τους τομείς δηλαδή είναι ιδιαίτερα ε, εκτεθειμένοι, όπως για παράδειγμα οι Βαλτικέ χώρες και ίσως και η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Κατά τα άλλα όμως οι χώρες μέλη βρίσκονται σε συγκρίσιμη θέση και με την Ευρωζώνη. Ενδιαφέρον στο γράφημα αυτό είναι ότι η έκθεση στον κίνδυνο των συναλλαγματικών ισοτιμιών για παράδειγμα για χώρες όπου ο τραπεζικός τομέας είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας όπως η Τσεχία και η Σλοβακία παρόλα αυτά έχουν θετική ε, θέση του τραπεζικού του τομέα σε σχέση με ε, τις διακινήσεις κεφαλαίων από την Ολοδαπή. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πια ότι η έκθεση στις ε, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών εξαρτάται από τη διαχείριση του τραπεζικού τομέα, από τη διαχείριση των τραπεζών. Στις χώρες λοιπόν μέλη, ανεξαρτήτως αν είναι παλές ή που έχουν ωστόσο υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και πολιτικές πίστης έχουν λιγότερη τάση να χρώνονται στην αλλοδαπή, να έχουν εξωτερικό χρέος δηλαδή και λιγότερη έκθεση σε δάνεια από το εξωτερικό και αυτές οι χώρες τα έχουν πάει καλύτερα στην κρίση. Και αυτό που τις βοήθησε επίσης ήταν και μια υγιής διαχείριση του τραπεζικού του τομέα είτε ήταν εγχώριας ιδιοκτησίας τράπεζες αυτές, είτε ήταν αλλοδαπής ιδιοκτησίας. Αντίθετα με χώρες όπου υπήρχαν συστημικές αδυναμίες, με μεγάλες εκθέσεις και όπου και η τιμή της στέγης για παράδειγμα. Ή χώρες οι οποίες είχαν ε, Παραδοσιακού τραπεζικού τομεί με παραδοσιακέ δραστηριότητε των τραπεζών κατάφεραν να ξεπεράσουν καλύτερα την κρίση ή να πληγούν λιγότερο. Το τρίτο μήνυμα είναι ότι εξακολουθούμε να έχουμε προκλήσεις μπροστά μας. Τα θέματα πολιτικής που δεν μπορούν να λυθούν εύκολα διότι έχουν πολύπλοκες είναι πολύπλοκα θέματα πολιτικής και θα παραμείνουν δύσκολα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρώτη πρόκληση είναι πώς να αντιμετωπίσουμε να υπάρξουν, να συσσωρευθούν ε, σημαντικές εξωτερικές επιβαρύνσεις για τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν άκαμπτες ή συναγματικές και αυτά τα προβλήματα είναι πολύ δύσκολο να επιληθούν. Η δεύτερη πρόκληση είναι πώς να εσωτερικοποιηθούν οι συστημικοί κίνδυνοι και να ενταχθούν στην διαχείριση κινδύνου που διεξάγουν οι τράπεζες. Και αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξει η τραπεζική εποπτεία, η εποπτεία του τραπεζικού τομέα. Να συνεννοηθεί με τις τράπεζες, να του ζητήσει να εντάξουν τον συστημικό κίνδυνο στο risk management που κάνουν, στα συστήματα διαχείρισης κινδύνου δηλαδή, ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να μην γίνουν εν τέλει κίνδυνοι της πίστης. Λόγω των προβλημάτων αξιοπιστίας είναι σημαντικό να υπάρξουν μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορέσουν να μειώσουν τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από ένα πανικό του κοινού που θα τρέξει στις τράπεζες να αποσύρει τα χρήματά του. Το ίδιο και για τους χρήστες του ευρώ για να αυξηθεί η αξιοπιστία του συστήματος. Και τέλος, αλλά σημαντικό, τα πακέτα δημοσιονομικής διάσωσης. Οι χώρες εκείνες οι οποίες διέσωσαν τους τραπεζικούς τους τομείς δηλαδή ή που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ύφεση με τεράστιες ενέσεις ε, ρευστό θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αργότερα και κυρίως οι χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στη ζώνη ευρώ, αυτό μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγάλη πρόκληση στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σμίτκοβα. Ο κύριος Ντάρκας τώρα θα μας παρουσιάσει τις δικές του απόψεις για τις ε, γενικές μακροπρόπτικες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν οι δύο προλογιστέντες ομιλητές. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που ακούσατε ήδη και να τονίσω διαφορετικές πτυχές. Καταρχήν, όπως είπαν και οι δύο μιλητές, χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπληρωμένων και των νέων πλήγησαν ε, πλήξαν πιο σκληρά από την κρίση. Τα χειρότερα προβλήματα των περασμένων κρίσεων όπως ε, προβλήματα με νομισματικά <coughs> και παραδείγματος χάρη είναι κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος κλπ. Η Όπως είπαν οι περισσότεροι που έδειξαν κάποια στοιχεία για το ΑΕΠ και πως το ΑΕΠ ε, μειώθηκε στις περισσότερες χώρες από την Πολωνία. Εγώ έχω ένα διαφορετικό στοιχείο για να το καταδείξω. Δηλαδή να δούμε πώς, ποια είναι η διαφορά της ανάπτυξης πριν από την κρίση και μετά την κρίση τι είναι η πραγματική επίπτωση της κρίσης, παραδείγματο χάρη. Αν κάποιος έχει μια ε, θέση απασχόλησης και έχει κάποιο εισόδημα, υπολογίζει ότι θα έχει το εισόδημα αυτό και στο μέλλον, ξαφνικά είναι άνεργος και παίρνει ε, επίδομα ανεργίας και επίσης τιμές αυξάνονται, άρα το διαθέσιμο του ε, εισόδημα είναι πολύ μικρότερο. Ο επόμενος πίνακας δείχνει Ε, την, ε, τα ποσοστά αυτά από την κρίση, κάπως διαφορετικά από εκείνα που είχαμε, σε όλες τις περιπτώσεις. Και συμφωνώ με την κυρία Σμιτκοβά. Σχετικά με όσα είπε για το Διεθνές Αμπισμότικο Τομείο. Αναφέρθηκε επίσης και ότι πολλοί από τους αναλυτές των αγορών συνενώνουν σε αυτές τις τράπεζες, εδώ βλέπετε, με μπλε χρώμα τις ε, παλιές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόκκινο είναι άλλες χώρες και κίτρινο είναι οι νέες χώρες μέλη. Οι άλλες χώρες, οι περιοχές της χώρας μου είναι Αφρική, Ασία, ε, Λατινική Αμερική κλπ. Βλέπετε ότι πάνω πάνω βρίσκονται οι τρεις ε, νέες χώρες ε, Λετωνία, Λιθουανία και Εσθονία, που επλήγησαν το περισσότερο όπως το είπαν και άλλοι. Μειώθηκε το ΑΕΠ τους κατά 30-40%. Τόσο πάρα πολύ σημαντικά δηλαδή. Μετά έχουμε τα άλλα νέα κράτη-μέλη με τρεις εξαιρέσεις. Την Κύπρο και την Μάλτα που είναι νέες χώρες βέβαια και τα προβλήματά τους δεν είναι τόσο μεγάλα. και η Πολωνία επίσης ως εξαίρεση. Αλλά οπωσδήποτε έχουν πληγεί περισσότερο νέες μέλη. Και γιατί υπάρχουν αυτές οι σημαντικές αλλά διαφορετικές επιπτώσεις. Καταρχήν, η ισχυρή ε, βάση πάνω στο σε κεφάλαιο έχετε εδώ ένα πίνακα που λέει πως η ροές του κεφαλαίου πήγαν στην Ανατολική Κεντρική Ευρώπη. Έχετε άμεσες ε, επενδύσεις, επενδύσεις χαρτοφυλακίου και άλλες ροές. Και βλέπουμε ότι ε, από το 2000 υπάρχει σημαντική αύξηση του κεφαλαίου, φτάνει στο 10% του ΑΕΠ για το σύνολο της περιφέρειας, που είναι πάρα πολύ μεγάλο, και ξαφνικά μειώθηκε στο 0. περάσου δεν υπήρχε έξοδος κεφαλαίου, ίσως εξαίρεση μικρές ποσότητες στην Λετωνία, αλλά ξακάθαρα δείχνει αυτή η εικόνα ότι υπήρχε σημαντική εισρωή κεφαλαίου που σταμάτησε. Γιατί, ποιοι ήταν οι λόγοι για την εισρωή του κεφαλαίου και ποιοι ήταν οι λόγοι για την ξαφνική διακοπή τους πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν εδώ οι εσωτερικές πολιτικές στις ε, τρεις χώρες της Βαλτικής. Παραδείγματος χάρη. Ε, είχατε, είχαν ένα σύστημα μέχρι την, ε, τις αρχές δεκαετίας του 2000 που δεν τροποποίησανε. Οι επιπτώσεις στην αγορά κινήτων ήταν αρνητικές και γι' αυτό αυξήθηκαν οι τιμές ε, και η ίδια μου χώρα, η Ουγγαρία, έκανε σημαντικότατα σφάλματα όσον αφορά την φορολογική της και η οικονομική της πολιτική. Ήδη σε μια περίοδο κατά την οποία η ε, ε, οικονομία στην Ευρώπη πήγαινε πάρα πολύ καλά, η Ουγγρική κυβέρνηση είχε σημαντικότατα ελλείμματα. Αυτό που θέλω κύριος να πω είναι ότι αυτή καθ' η ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντική, ε, σημαντικός παράγοντας αύξησης της ροής κεφαλαίων. Αν προσπαθήσει κανένας να δει δηλαδή ποιους άλλους λόγους μπορούμε να βρούμε που εξηγούν το ότι οι περιοχές αυτές βασίζονται στην ισορροή των κεφαλαίων. Υπάρχουν, όπως σας είπα, θέματα εσωτερικής πολιτικής, αλλά επίσης το θέμα της ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της έναρξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομική ολοκλήρωση εμπορική επίσης, που ήταν προς όφελος των χωρών, αλλά οδήγησαν και στα προβλήματα που γνωρίζουν σήμερα. Είναι αυτό. Δεύτερο. Το εμπόριο είναι πάρα πολύ σημαντικό στις χώρες αυτές. Και ορισμένες χώρες όπως η Σλοβακία, παραδείγματος χάρη, είχαν εξαγωγές στον τομέα της αυτογενομηχανίας, μια βιομηχανία που επλήγει περισσότερο από την κρίση και γι' αυτό η Σλοβακία επλήγει επίσημα από την κρίση. Επίσης, πολλές από αυτές τις χώρες Ε, είχαν στο παρελθόν πολλές αποστολές χρημάτων από μετανάστες σε άλλες χώρες που μειώθηκαν. Γιατί η κατάσταση στην Δυτική Ευρώπη είχε αυτή την επίπτωση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αναφέρθηκα στις ευθύνες που υπάρχουν για το πόσο ευάλωτες ήταν οι οικονομίες αυτές που Επίσης μπορώ να συμφωνήσω ότι η Ανατολική Ευρώπη ή οι τέλο πάντων οι χώρες μέλη αυτή δεν είναι ομοιογενής ε, ομάδα. Υπάρχουν δύο τουλάχιστον υποδομάδες και μπορώ να συμφωνήσω με προλέσσαντες ότι υπήρχαν σημαντικότητε αλλαγές όσον αφορά το τα εμπορικά για των δύο χρόνων αυτών. Γιατί είχαν 5, 6, 7% έλλειμμα ε, ισοζυγίου, αλλά για τις εξαγωγές, εισαγωγές υπήρχε μία ισορροπία. Και μάλιστα, άμα δούμε τώρα άλλες χώρες, χώρες Βαλτικής, Βουλγαρία, Ρουμανία, δούμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου. Η κατάσταση που υπήρχε δηλαδή δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και μπορώ να πω ότι οι περισσότερες χώρες βασιζόταν μέσα σε εισβολές κεφαλαίου, αλλά είχαν κάποια βασιμότητα, ενώ οι χώρες της ε, Βαλτικής και η Βουλγαρία και η Ρουμανία όχι. Πώς μπορέσουν να αποφευθούν τα χειρότερα προβλήματα των παλαιών κρίσεων Καταρχήν υπήρχε πάρα πολύ έντονη αντίδραση του διεθνού κοινότητα με παραδείγματο του δάνεια προς τις τρεις χώρες αυτές. Επίσης ε, δόθηκαν χρήματα εκ των προτέρων από τα ταμεία, τα διαφορετικά και το Ταμείο Συνοχής, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επινοικοδόμησης. Όλα αυτά ωφέλησαν προφανώς τις χώρες που δέχτηκαν τα λόγο κεφάλαια. Επίσης, ο τραπεζικός τομέας ήταν πολύ πιο σταθερός, λιγότερο ευάλωτος από ότι σχετικά με άλλες κρίσεις όπως την κρίση της Ασίας. Επίσης, εξωτερικές ε, ήθοι οι αλλοδαπές τράπεζες, συγγνώμη, παρέμειναν δεσμευμένες στην περιφέρεια αυτή. Η πρωτοβουλία αυτή της Βιέννης, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που βοήθησε τις ε, χώρες αυτές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέθεσε ρευστό χρήμα και επίσης υπήρχε και μια πολιτική δέσμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηριχτούν ε, πολλά έγιναν πολλά καλά έγιναν θα έλεγα. Εγώ είμαι πολίτης μιας νέας χώρας μέλους και πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τη βοήθεια που εδόθηκε και στη χώρα μου. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά και κάποιοι κίνδυνοι. Ο, φόρος, ο ρόλος των εξωτερικών τραπεζών, των αδραπών τραπεζών, που ήταν πάρα πολύ σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη πριν από την κρίση. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. βοήθησε τι χώρε αυτέ να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό τραπεζικό σύστημα που ήταν πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά όμως συνέβαλαν στο ευάλωτο των χωρών αυτών πριν από την κρίση. Η Κατερίνα έδειξε κάποιε διαφάνειες για το ε, ποιες επιπτώσεις υπήρχαν ε, όσον αφορά την τιμή των ακινήτων. Τα ακινήτα αυξάνονται κατά 5% έτος δεν μπορεί να μας εκπλήξει ότι αυτή η φούσκα κάποια στιγμή έσκασε στην Λετωνία Φιλιππίν. Οι ε, τιμές των ακινήτων έπεσαν κατά 70% το 2 τρίτο, δηλαδή της αξία τους χάθηκε. Και πάλι ο λόγος για την ε, τίναξη αυτή της αγοράς ακινήτων οφείλ, ήταν εν μέρη ε, και οφειλόμενος στην, ε, στην δραστηριότητα των ε, αλλοδαπών τραπεζών στις χώρες αυτές. Όσον αφορά το μέλλον, είμαι πάρα πολύ ε, επιφυλακτικός ότι θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ε, νέες χώρες μέλη όταν οι τράπεζες αρχίσουν ε, να κάνουν τις απαραίτητες μετατροπές που χρειάζονται. Ε, ιδίως αν αποσυρθούν, ακόμα και αν δεν αποσυρθούν, από ό,τι ακούσαμε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αποσυρθούν, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα δίνονται επαρκή σε επιστώσεις στο μέλλον. Ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως είπα, είχε δώσει μια άμεση ενίσχυση. Ήταν όμως εκπληκτικό ότι έδωσε συμφωνίες swap στην Δανία και στη Σουηδία, δύο χώρες που είναι εκτός του χώρου ευρώ, χωρίς να δώσουν τίποτα παρόμοιο σε άλλες χώρες. Από ό,τι ξέρω, η Πολωνία, η Λετωνία υπάρχουν διαφορές και είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε. Δεν θα τα αναφέρω όλα αυτά τώρα. Θα σας πω κάτι σχετικά με τις επιπτώσεις κρίσης στο μέλλον. Μία κύρια εξαίρεση είναι η Εσθομία που θα ζητήσει να ενταχθεί φέτος. Το ΕΠ ε, κατέρευσε κατά 20% σε δύο χρόνια. Ξέρετε, ο περισσότερο ήταν κάτω από το 30%. Η Εστονία όμως ε, παρόλη την μείωση αυτή του ΕΠ έμεινε στο 3% του χρέους. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ αξιόλογη αυτή η συμπεριφορά αυτής της χώρας και γι' αυτό κατά πάσα μενότητα η αίτηση της Εστονίας θα γίνει δεχτή. Παρ' όλα αυτά προβλέπεται βέβαια ένα κριτήριο αηφορίας, το οποίο δεν είναι πολύ ακριβό στη διατύπωσή του και δεν ξέρουμε η Κομισιόν και η Κεντρική Τράπεζα όταν εξτάσουν το, την έκθεση σύγκρισης πώς θα το εκτιμήσουν αυτό. Ελπίζουμε πραγματικά ότι η Εστονία θα καταφέρει να ενταχθεί. Για όλες τις ε, άλλες χώρες όμως η πιθανότητες να ενταχθούν στο ευρώ έχουν μειωθεί σημαντικότατα. Λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ελλανδία, η Ελλάδα πραγματικά ε, είναι μια μεγάλη δοκιμασία γιατί κανένας δεν περίμενε ότι ένα κράτος μέλος τους Ευρωζώνης θα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση. όλα τα νέα κράτη-μέλη, εξαίρεση πάντα τη Ουγγαρία, είναι πολύ διαφορετικέ από την Ελλάδα όσον αφορά τη φορολογική του πολιτική. Το ε, χρέος παραδείγματο χάρη είναι 7% στην ιστορία του, στην, ε, του ΑΕΠ στην Ουγγαρία, συγγνώμη. Είναι πολύ πιο υγιεί οι χώρε αυτές λοιπόν από την Ελλάδα. Ένα σημαντικό θέμα είναι κατά πόσο πρόκειται να ενταχθούν νέα μέλη στην Ευρωζώνη. Γιατί οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα, στην Ισπανία, μειώνουν την τάση για την πρόσκληση νέων χωρών μελών στην Ευρωζώνη. Είναι περίεργο επίσης ότι το 2010-2011 κανένα από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης θα πληρούν όλα τα κριτήρια. Αλλά οι χώρες που είναι υποψήφιες και ζητούν να ενταχθούν πρέπει να εκπληρούν όλα τα κριτήρια αυτά. Περίεργο μου φαίνεται. Λοιπόν, το θέμα της ευρώ είναι σημαντικό. Ορισμένες χώρες έχουν αρκετά ευέλικτες οικονομίες και έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν. Άλλες χώρες, όπως η Πολωνία και η Τσεχία, ίσως δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ να ενταχθούν. αλλά φοβούμαι ότι πραγματικά η κρίση μειώνει σημαντικά τις ε, δυνατότητες των χωρών να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Σας ευχαριστούμε κύριε, κύριε Ντάρβας. Έχουμε προβλέψει περίπου μία ώρα για ερωταπαντήσεις. Θα ακούμε τρεις ερωτήσεις και μετά θα δίνουμε το λόγο στους καλεσμένους μας για απαντήσεις. Ο κύριος Στόλογιαν, παρακαλώ να πείτε σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω ερώτηση προς τον κύριο Κέρεμανς. Γνωρίζετε ότι η Ρουμανία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τον όρο να απελευθερωθούν τα οι κεφαλικοί λογαριασμοί. Αυτή ήταν προϋπόθεση για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο είδαμε μια ηλικιώδη αύξηση του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέους. Και αυτό το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος ευνοήθηκε από τις ε, τράπεζες και τις ε, πολυεθνικές εταιρείες και μάλιστα πριν την κρίση αυτό το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος ισοδυναμούσε περίπου στις στα διεθνή αποθέματα της Ρουμανίας, στα αποθέματα σε διεθνή συναλλάγματα. Παρόμοια κατάσταση αντιμετώπιζε η Νότια Κορέα πριν αντιμετωπίσει κρίση. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τάση αύξησης του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέους. Και τότε θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για να αναχαιτιστεί αυτή η αρνητική τάση του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέου που στην περίπτωση τη Ρουμανία δημιούργησε τεράστιο κίνδυνο και μπλοκαρίστηκε εξαιτία τη υποχρέωση που είχε αναλάβει για την ένταξη. Ποια είναι η δική σα γνώμη, κυρία Μπέρε. Όχι, δεν έχει ερώτηση. Η κυρία Γιώρη. Σας ευχαριστώ στα Ουγγρικά. Σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μας δίνετε για συζήτηση και ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους. Ευχαριστώ την κυρία Σμίτκοβα για τις ε, πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που υπέβαλε. Φυσικά δεν επιτρέπονται οι γενικεύσεις και δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα μέλη της Ευρωζώνης παρόμοια με τις χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Και αν υπάρχει ένα δίδαγμα που μπορούμε να αντλήσουμε, είναι ότι η κυβερνητική πολιτική μιας χώρας καθορίζει την κατάσταση της χώρας αυτής, άσχετα από την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί κάθε χώρα, ανάλογα με την κυβερνητική πολιτική που ακολουθεί, μπαίνει και σε συγκεκριμένο δρόμο. Ας μην γενικεύουμε λοιπόν και να κρίνουμε αξιοκρατικά κάθε χώρα ανάλογα με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα που υποβάλλει. Υπάρχουν πολλά συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε. Διαπιστώνουμε ότι οι μικρές χώρες με ανοιχτές οικονομίες, δεν είναι βέβαια μικρές μόνο οι χώρες, γιατί η Πολωνία είναι αρκετά μεγάλη χώρα, αλλά οι χώρες που εξαρτώνται σε αλλοδαπή χρηματοδότηση είναι και πιο ευάλωτες εξαιτίας του ότι βρίσκονται εκτός ευρωζώνης. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Γιατί οι χώρες που προσχώρησαν, που εντάχθηκαν στην Ένωση το 2004, ανέλαβαν την υποχρέωση να ενταχθούν αργά ή γρήγορα στην Ευρωζώνη και άρα υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν οικονομικές πολιτικές με απότερο στόχο την προσχώρησή τους στην Ευρωζώνη. Και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε η πρόθεση θεσμοθέτησης της Ευρωζώνης και πιο αυστηρής περιχαράκωσής της. Αυτό προβλέπει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Πάντως προσοχή, θα ήθελα να σας κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου γιατί Κάτι τέτοιο θα ορθώσει πολύ πιο ανυπέρβλητα εμπόδια για ένταξη των νέων χωρών. Ποια είναι η δική σας γνώμη γι' αυτό. Γιατί εγώ διαπιστώνω μια αντίφαση. Η τρίτη παρατήρησή μου αφορά την ευθύνη των κυβερνήσεων. Πολλοί εστιάζονται τελευταία στην περίπτωση της Ελλάδας, αλλά ο κύριος Ντάρβας ανέφερε ότι η Ουγγαρία ήταν χαρακτηριστική περίπτωση. αποδεικνύει ότι αν κανείς προσπαθεί να θολώσει τα νερά με τα στοιχεία και δεν υποβάλει ακριβή στοιχεία, αργά ή γρήγορα θα ξεμπροστιαστεί. Βέβαια το πρόβλημα τώρα δεν είναι η Ουγγαρία αλλά η Ελλάδα. Είναι προφανές πάντως ότι όταν μια χώρα, μια κυβέρνηση δεν δίνει ακριβή στοιχεία, ε, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Όσο πιο ακριβή στοιχεία υποβάλλει, τόσο πιο ξεκάθαρε πολιτικέ μπορεί να ακολουθήσει. Η Πολωνία, παρόλο που αντιμετώπισε και αυτή η κρίση, διαφύλαξε μια θετική οικονομική ανάπτυξη και στην διάρκεια της κρίσης. Οι χώρες της σύγκλησης κατάφεραν να αποφύγουν τους χαλεπότερους ε, καιρούς της κρίσης. θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν φαίνεται ποιες χώρες αξιοποίησαν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάκαμψης. Η Ουγγαρία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε όλα τα κονδύλια, πήγε ε, στο κόκκινο του λογαριασμού της, ισόρευσε χρέος και στην περίοδο των παχιών αγελάδων και όταν ε, χτυπήθηκε από την κρίση δεν κατάφερε να ορθοποδήσει δεν, μπορούσε, δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τις συστάσεις του σχεδίου ανάκαμψης, ούτε να αξιοποιήσει τα κονδύλια που στόχο είχαν την ε, αναζωγόνηση της οικονομίας. Και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Και ακόμη και φέτος η Ουγγαρία θα παρουσιάσει αρνητική οικονομική ανάπτυξη, γιατί δεν κατάφερε ακόμη να αναζωογονήσει την οικονομία της. Γιατί είχε εξαντλήσει πριν καν να αρχίσει η κρίση τα αποθέματά της. Μία άλλη παρατήρηση για τις δραστηριότητες των αλλοδαπών τραπεζών. Κανένας δεν αμφιβάλλει για την ανάγκη δραστηριοποίηση αυτών των αλλοδαπών τραπεζών που συμβάλλουν τα μάλα στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά ακόμη και σε ένα μήνα μπόρεσαν να απομακρύνουν 3 δις ε, ευρώ από την Ουγγαρία και μόνο. οι αλλοδαπέ τράπεζε μπορεί μερικές φορές να επιτείνουν τον ευάλωτο χαρακτήρα των οικονομιών αυτών των χωρών. Θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει νέους ε, χρηματοπιστωτικούς και δημοσιονομικούς κανονισμούς. Λαμβάνεται υπόψη τη επιπτώση των νέων δημοσιονομικών κανονισμών στι νέε χώρε μέλη. Αν αυξηθούν οι κεφαλαϊκέ ανάγκες των τραπεζών, οι τράπεζε αυτέ που δεν έλαβαν ε, έχεις κεφαλαίου, νέες κεφαλαίου, όπως οι τράπεζες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, θα έρθουν σε δυσμενή θέση και σε λιγότερο ανταγωνιστική θέση, γιατί θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις κεφαλαιακές τους υποχρεώσεις και να αυξήσουν τα κεφαλαία τους, κάτι που θα τους οδηγήσει να περικόψουν τα δάνεια που δίνουν. Με αποτέλεσμα να πληγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές και στις χώρες αυτές. Μπορείτε να εκτιμήσετε τις επιπτώσεις της εφαρμογής του νέου δημοσιονομικού κανονισμού στις νέες χώρες. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι στις ερωτήσεις για να προλάβουν όλοι να τις θέσουν. Κυρία Χιούμπνερ είναι η τελευταία ομιλήτρια σε αυτό το γύρο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τον τραπεζικό κλάδο ο κύριος Κέρεμανς, αν δεν κάνω λάθος, ε, υπέβαλε τα σχετικά σχόλια και τον ρωτώ, μετά τις εκτενείς αναλύσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς πιστεύετε ότι υπονόμευσε η κρίση τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια. Πώς επηρέασε η κρίση τα ισοζύγια πληρωμών των τραπεζών, τους ισολογισμούς των τραπεζών στις νέες χώρες μέλη. Και αυτό υπό το φως ε, της ανασυγκρεώτησης, ε, επανειδιωτικοποίησης, επανακεφαλαιοποίησης. Πώς θα επηρεαστεί από, τα, από τις νέες απαιτήσεις ο τραπεζικός κλάδος, ιδιαίτερα στις νέες χώρες. Κυρία Σμίτκοβα, αν συγκρίνετε τις χώρες που έχουν ε, σχετικά άκαμπτη ισοτιμία με αυτές που έχουν κειμενόμενη, βλέπετε ότι αυτές με την άκαμπτη είναι πιο ευάλωτες. Μπορείτε να συγκρίνετε την κατάσταση μεταξύ χωρών Ευρωζώνης και χωρών εκτός Ευρωζώνης. Τι επίπτωση θα είχε η συμμετοχή στην Ευρωζώνη σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα ή την ανθεκτικότητα ή τη δυνατότητα επαναφοράς μετά από μια κρίση. Κύριε μας νομίζω ότι προς εσάς σας απευθύνονταν οι περισσότερες ερωτήσεις, οπότε θα ξεκινήσουμε με εσάς. Καλώ, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που τις ακούσαμε. Πρώτη ερώτηση από τον ε, Ρουμάνο Ευρωβουλευτή για την περίπτωση της Ρουμανίας και την ε, ξαφνική έλλειψη ισορροής κεφαλαίων. και ε, η επίπτωση από την προσήλωση στο φετίχ της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. Πολύ εύστοχη ερώτησή σας, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σκέφτηκε μερικές φορές την πιθανότητα ε, διενέργειας ε, βραχυπρόθεσμου κεφαλαικών ελέγχων για να αποφευθούν κερδοσκοπικές εισρωές κεφαλαίων. Τελικά όμως ε, δεν τελεσφόρησε αυτή η πρόταση για τέτοιους ελέγχους. Καταρχήν γιατί μπορεί εύκολα κανείς να παρακάμψει τέτοιους ελέγχους και ήταν ένας από τους λόγους που απέτρεψαν τη θέσπισή τους. Και μερικές φορές όταν υπάρχουν ε, ενδείξεις για προβλήματα ανεπίλητα σε μια χώρα, συνήθως λαμβάνονται πιο ορθόδοξα μέτρα που ευθυγραμμίζονται με την οικονομία της αγοράς και αποφεύγονται μέτρα που στρεβλώνουν μια ομαλή λειτουργία της αγοράς για να αποφευθεί εκτροπή των κονδύλιων των πόρων όταν ε, εφαρμοστούν αυστηρή ελέγχοι κεφαλαίου. Τώρα, ποια είναι η εναλλακτική λύση. Πολύ συχνά νομισματική πολιτική δεν είναι και πολύ αποτελεσματική, γιατί μαζικές ισορροές κεφαλαίων ε, συνοδεύονται από πληθωρισμό, από αύξηση επιτοκίων, από ακόμη μεγαλύτερη διόγκωση της ροής, κάτι που δεν βοηθάει. Το, αυτό που βοηθάει περισσότερο είναι μια πιο αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, κάτι που προϋποθέτει ε, κακά μαντάτα προς τους ψηφοφόρους και αυτό δεν ικανοποιεί ιδιαίτερα τους πολιτικούς, γιατί φοβούνται την, ε, το boomerang από την αντίδραση των ψηφοφόρων τους. Οπότε αποφεύγει κανείς τους ελέγχους κεφαλαίων και σε πολλές χώρες μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική παρόλο που χρειαζόταν δεν εφαρμόστηκε. Και γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε επιδείνωση της κατάστασης. Αυτός προς την πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση υπευλήθη από εκπρόσωπο της Τσεχίας. Δεν ξέρω αν ήταν από την Τσεχία η κυρία. Α, συγγνώμη, από την Ουγγαρία ήταν η Ευρωβουλευτής που υπέβαλε τη δεύτερη ερώτηση. Εγώ αγγλικά άκουγα, γι' αυτό δεν μπόρεσα να καταλάβω αν είσαι από τη Τσεχία ή από την Ουγγαρία. Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, ρωτήστε ποια είναι η επίπτωση του, των νέων δημοσιονομικών κανονισμών που εκπονούνται στις τράπεζες των νέων χωρών. Προτιμάτε πιο αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίου περισσότερες απαιτήσει ε, κεφαλαίου και άρα μεγαλύτερη δυσκολία εξαιτία της δύσκολης πρόσβασης στα δάνεια, ιδιαίτερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε όλοι ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτών των πιο αυστηρών διατάξεων των δημοσιονομικών κανονισμών και Πολλές φορές η δημοσιονομική κρίση διαβρύνθηκε εξαιτία της υπερβολικής κερδοσκοπίας, της υπερχρέωσης και αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν. Και αν θέλει κανείς αποφύγει ελέγχους κεφαλαίου, που πολλοί απέφχονται γιατί αντιβαίνουν στους, στην ελευθερία κυκλοφορίας, το μόνο μέτρο που μπορεί να θεσπιστεί είναι η μεγαλύτερη κεφαλαϊκή απέτηση από τις τράπεζες. Υποχρέωση αύξηση του κεφαλαίου. Βέβαια, οι περισσότερες χώρες ούτω ή άλλω τηρούν ε, τέτοιε απαιτήσει, γιατί οι αγορέ το απαιτούν. Συνήθω ε, κανονιστικά θα πρέπει να είναι πάνω από 8%. Οπότε πρέπει να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο για να ρυθμιστεί το τραπεζικό σύστημα. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εφαρμοστεί και όλα. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση οικονομική είναι παραπέουσα. Και εκεί θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία εξετάσαμε και το ρόλο της ε, ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ε, αποκατέστησε μια ρευστότητα στην οικονομία, γιατί υπήρχε δυσπιστία μεταξύ των τραπεζών και χρειάστηκε επέμβαση ε, με ισορροή κεφαλαίων από την ΕΚΤ. Αυτά τα χρήματα όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να τα απορροφήσει πίσω, να τα απο... η ΕΚΤ. Βέβαια, αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν ε, για δάνεια και αυτή τη στιγμή λόγω συρρήκνωσης της οικονομίας δεν υπάρχει, απέ, δεν υπάρχει αίτηση, ζήτηση δανείων. Κάπως όμως θα πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομία. Και η κυρία Χιούμπνερ, <laughs> Πολωνέζα, είμαι σίγουρη για την καταγωγή της, γιατί ήσασταν και πρώην επίτροπος αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αναγνώρισα από πού είστε. Το θέμα της ε, αναδιάρθρωσης των τραπεζών. και της κατάστασης εκεί. Είναι περισσότερο θέμα ανταγωνισμού. Γιατί κάποιες τράπεζες έλαβαν πολλές κρατικές ενίσχυσεις, πολλά κονδύλια από το κράτος, όχι τόσο στην Πολωνία, γιατί ήταν από τις λίγες χώρες η Πολωνία που απέφυγε την κρατική επέμβαση. Αλλά σε άλλες χώρες, όπως η Λετωνία για παράδειγμα, στην Ουγγαρία δόθηκαν δαψιλός κονδύλια από το κράτος προς τις τράπεζες για να αποφευθεί όξυνση της κρίσης και μάλιστα υπήρξε ανάγκη και για διεθνή αρρωγή. Οι τράπεζες αυτές θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν και να περιορίσουν ίσως τις δραστηριότητες τους γιατί οι κρατικές ενισχύσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση των τραπεζών και του μεριδιού τους στην αγορά γιατί αυτό θα ήταν αθέμητος ανταγωνισμός προς τις άλλες τράπεζες. Οπότε στην αναδιάρθρωση και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων σε αυτές τις τράπεζες που έτυχαν της κρατικής ενίσχυσης, δεν μπορούμε να περιμένουμε συμβολή τους στην οικονομική ανάκαμψη. Πάντως ισχύει η γενική αρχή της ελεύθερης αγοράς και των όρων θεμητού και υγιούς ανταγωνισμού. Οπότε οι τράπεζες που έτυχαν κρατικής ενίσχυσης οφείλουν να αναδιαρθρωθούν και αυτή θα είναι χρονοβόρα διαδικασία. Επίση, θα πρέπει μέσα σε μία πενταετία να επιστρέψουν τα κρατικά κονδύλια που έλαβαν. Και αφού επιστρέψουν το χρέος τους, τότε μπορούν να, να διευρύνουν και πάλι τις δραστηριότητές τους. Αυτά ως προς ερωτήσεις που ήταν για μένα. Κυρία Σμίτκοβα. Πρώτα για το σχόλιο σχετικά με το μέγεθος της χώρας. Βέβαια, το μέγεθος της χώρας ήταν ένας από τους παράγοντες που δεν αναφέρθηκαν ρητά στην παρουσίαση. Βέβαια έχει σημασία από την άλλη μεριά η Σλοβακία και η Τσεχική Δημοκρατία που δεν είναι μεγάλες χώρες, είναι αρκετά μικρές και όμως τα κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κρίση σχετικά καλά. Υπάρχουν λοιπόν δύο παράγοντες που αναφέρθηκαν και από τους άλλους ομιλητές που έχουν μεγαλύτερη σημασία από το μέγεθος της χώρας. Εάν δηλαδή η χώρα είναι ικανή ή όχι να προσελκύσει επαρκείς ε, εγχώριες καταθέσεις για να χρηματοδοτηθούν τα δάνεια, τότε δεν έχει σημασία αν είναι μικρή, διότι δεν εξαρτάται από διαμεθοριακές κινήσεις κεφαλαίων και βέβαια και η εξοπιστία των εγχωρίων πολιτικών και η ιστορία των πολιτικών. Μπορεί να έχει ιστορία 50 ετών που δεν μπορεί να αλλάξει τόσο γρήγορα. Είναι λοιπόν και η ιστορική αφετηρία της κάθε χώρας, από που ξεκινά δηλαδή, αλλά και από τους άμεσους ε, στόχους των εξωτερικών επενδύσεων. Εάν δηλαδή πηγαίνουν περισσότερο στον εμπορικό τομέα, αναπτύσσουν τότε την εξαγωγική ικανότητα της οικονομίας, ακόμα και μια μικρή χώρα μπορεί τότε να παραγάγει επαρκές εισόδημα από τις εξαγωγές για να ε, χρηματοδοτήσει και τα δάνεια ή εάν πάει για παραδείγμα στην, ε, στα ακίνητα η επένδυση αυτή. Οπότε η κατάσταση δεν είναι το ίδιο καλή. Έχουμε στο δεύτερο σχόλιο που έχει σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών. Συχνά λέχθηκε ότι μια χώρα που μπαίνει στη ζώνη ευρώ το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών εξαφανίζεται. Όμως στις χώρες, στην ομάδα χωρών μελών με υψηλή εξωτερική χρέωση, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, παρόλο που στην επιφάνεια εκλείπουν ε, ε, ε, τα προβλήματα, παρόλα αυτά <clears throat> παραμένουν τα χρέη. Ας είναι σε ευρώ, πρέπει να αποπληρωθούν. Το ερώτημα λοιπόν εάν οι χώρες, μέλη, οι χώρες μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν το συντομότερο δυνατόν το ευρώ ώστε να αποφύγουν τέτοιες κρίσεις στο μέλλον δεν είμαι τόσο βεβαία ότι από μόνο του το ευρώ μπορεί να διασώσει τις χώρες από το βάρος της κρίσης αν δεν υπάρχουν υγιείς εγχώριες πολιτικές αλλά και σε κάποιο βαθμό και καλή τύχη. Δεν θεωρώ λοιπόν την υιοθέτηση του ευρώ ως τη μοναδική λύση για τη διάσωση των χωρών. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και τα προβλήματα αξιοπιστίας που όπως ε, είπα από αυτήν εξαρτάται και η δυνατότητα προσέλκυσης εγχωρίων αποταμιεύσεων για τη χρηματοδότηση των ε, ε, τραπεζών ώστε να αποφευθεί το πρόβλημα αξιοπιστίας που ίσως αυτό επιτρέπει να αποκατασταθεί ένα ισοζύγιο. Βρίσκω ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία οι παράγοντες αυτοί από ότι η επίσημη εκδοχή. Σε ό,τι αφορά το ρόλο των αλλοδαπών τραπεζών, σε μία διαφάνεια προσπάθησα να δείξω την έκθεση σε αλλοδαπά δάνεια δεν έχει το σημασία εάν είναι αλλοδαπή ιδιοκτησία ή εγχώρια ιδιοκτησία οι τράπεζε, γιατί ορισμένε χώρε δεν είναι εκτεθειμένε σε δάνεια τη αλλοδαπή, όπω η Τσεχική Δημοκρατία. Και ορισμένε έχουν έχουν εγχώριας ιδιοκτησία και τράπεζε και όμω είναι εξαρτημένε από αλλοδαπέ ε, εισρωέ κεφαλαίων. Άρα δεν θεωρώ ότι φταίνε οι αλλοδαπές τράπεζες για ε, την πρόκληση της κρίσης. Ε, εφόσον οι πολιτικές ήταν υγιείς, ε, θα βοηθούσαν τις χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση. Εξαρτάται δηλαδή και από το επίπεδο πώς γίνεται η διαχείριση των τραπεζών και αν μπορούν να εσωτερικοποιήσουν την διαχείριση του κινδύνου. Υπήρξε, ε, τέθηκε και μια ερώτηση σχετικά με το εάν οι νέοι κανόνες εποπτείας ενδέχεται να δημιουργήσουν επιπρόσθετα προβλήματα και ιδίω ε, σχετικά, η ανάγκη σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου. Στις χώρες όπου υπήρξε υγιής διαχείριση των τραπεζών, αλλά και υγιής εποπτεία των τραπεζών, οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να εξεύρουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Πάλι για παράδειγμα η τσεχική δημοκρατία όπου κάθε τρίμηνο κάνουμε ένα stress test στο τραπεζικό τομέα και αν δούμε ότι οι τράπεζες δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κάποια σοκ σε ό,τι αφορά την πτυτικότητα την ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τότε τους ζητούμε να αυξήσουν την κεφαλαιακή τους βάση ώστε λοιπόν εν τέλει έχουν ίσως και πλονασματική κεφαλαϊκή βάση. Αυτό μπορεί να γίνει σε ε, χώρες όπου είναι υγιής η εποπτεία των τραπεζών και αυτό είναι βέβαια και πρόκληση για τους υπευθύνους. Πρέπει να εποπτεύουν τις τράπεζες προσεκτικά, να κάνουν τα stress test σε τακτική βάση και να ζητούν από τις τράπεζες να προβαίνουν σε αύξηση του κεφαλαίου τους εφόσον υπάρχουν ε, υπάρχουν, ε, ε, εφόσον διαγράφονται στο μέλλον προβλήματα. Και βέβαια, στις δύο ομάδες οι μηχανισμοί προσαρμογής είναι παρόμοιοι. Και αν ε, δεν υπάρχει επαρκή ευκαμψία στην οικονομία, στην αγορά εργασίας, γιατί τότε χώρες και στις δύο ομάδες πλήττονται με τον ίδιο τρόπο. Θα αυξηθεί το εξωτερικό τους χρέος, θα επιβραδύνει η οικονομία τους, αλλά επειδή και προηγουμένως μίλησα για την αξιοπιστία, οι χώρες μέλη της ζώνης ευρώ αντιμετωπίζουν καλύτερα τα προβλήματα, διότι είναι πιο αξιόπιστες και έχουν και τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν credibility schemes της ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επομένω μπορούν να αποκρούσουν κάπω καλύτερα την κρίση. Πάλι λοιπόν, από την άποψη αυτή, εάν έχουν ακολουθήσει υγιείς οικονομικές πολιτικές, έχουν μάλλον και καλύτερες βάσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την κρίση. Εσείς κύριε Νταρβάς. Θα επανέλθω σε κάτι που αναφέρε η κυρία Ντουρίας. Αλλά εδώ διαφωνώ λίγο. Δεν είναι μοναχα η ελληνική κρίση που οφείλεται σε δημοσιονομική ανευθυνότητα. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία όπου υπήρξε ένα boom στη στέγη και όμως αντιμετώπισαν βαρύτερα προβλήματα γιατί μετά από το σκάσιμο της φούσκας στην στέγη ε, πλήττονται πολύ βαριά οι χώρες αυτές ενώ στις καλές εποχές υπήρχαν και φορολογικά κίνητρα για παράδειγμα στην Ισπανία για τον τομέα του ακινήτου επομένως και οι εγχώριες πολιτικές ζήτησης ε, συνέβαλαν Στο επίπεδο της ζώνης ευρώ υπάρχουν κάποιες συμφωνίες. Συμφωνώ όμως με την ιδέα ότι η άσκηση πολιτικής στην ζώνη ευρώ, η άσκηση οι πολιτικών μέσα στην ζώνη ευρώ θα πρέπει να προσεγγίσει ε, και βέβαια συμφωνώ μαζί σας στο εξής δεν θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να πλήξει νέες χώρες που θέλουν να εισέλθουν στην ζώνη ευρώ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο τρόπος με τον οποίο παρέσχε ρευστότητα, μείωσε για παράδειγμα την ποιότητα των μηχανισμών που δέχθηκε για την αναχρηματοδότηση, άρα αυτό σήμαινε ότι όλοι οι μηχανισμοί εκείνοι οι οποίοι κανονικά δεν ήταν επιλέξιμοι, παρόλα αυτά εφαρμόστηκαν. Δεν αναφέρθηκα στην Ουγγαρία, αναφέρθηκα στην Πολωνία, η πολωνική κυβέρνηση η οποία υπέστη σοβαρά πλήγματα στη διάρκεια της κρίσης, αλλά παρόλα αυτά είχε ασκήσει πολύ υπεύθυνη πολιτική την προηγούμενη δεκαετία. Παρόλα αυτά υπήρξε πανικός μεταξύ των Πολωνών υπευθύνων, όπου από το 3 ε, περίπου φτάσανε στο 5% απέναντι στο ευρώ και εκεί αυτό προκάλεσε πανικό στην Πολωνία. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να δεχθεί ως επιλέξιμα τα πολωνικά κρατικά ομόλογα σε σλότη για αναχρηματοδότηση από την Τράπεζα Ευρώ. Αν υπάρξει όμως κάποιο συντονισμό πολιτικής, κάποιες διευκολύνσεις μπορούν να υπάρξουν για τις ε, νέες χώρες μέλη που αποδίδουν καλά όπως η Πολωνία και να ληφθούν κάποια μέτρα ώστε να μην ε, βλαβούν οι χώρες αυτές στη διάρκεια της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτός από τα ονόματα που προανέφερα, υπάρχει κανείς άλλος που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Τότε θα κλείσουμε τον ε, κατάλογο των ομιλητών και θα δώσουμε πρώτο λόγο στην κυρία Γιακονσάρη. Ωραία, ευχαριστώ. Ακούσαμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων χωρών μελών. Ερώτηση. Μπορείτε να πείτε λίγο περισσότερα σχετικά με τον πολιτικό πολιτισμό της κάθε χώρας. Υπάρχουν παραδείγματα από χώρες οι οποίες μπόρεσαν να επιλύσουν και τέλος πάντων να ξεπεράσουν τα προβλήματα της κρίσης. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των χωρών εκείνων οι οποίες προσπαθούν να επιτύχουν συνένεση στο πολιτικό επίπεδο και απέναντι στις χώρες εκείνες οι οποίες είναι πιο πολύ όπως Αμερική η οποία έχει πιο έντονες πολιτικές διαμάχες ποιες έχουν την καλύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και επίσης είπατε συχνά ότι η Πολωνία είναι καλό παράδειγμα αντιμετώπισης της κρίσης. Μπορείτε να πείτε λίγο περισσότερο, λίγα περισσότερα λόγια για την υπόθεση της Πολωνίας που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Κάλβιν. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Γιατί σε ορισμένα σημεία διαφωνώ με του ε, εκπροσώπου του εμπειρογνώμενου. Καταρχήν, θα πρέπει να μιλήσουμε με το δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου αυτού, που δεν είναι μια αντιπαράθεση παλιών και νέων κρατών, αλλά το επίπεδο της ε, οικονομικής ανάπτυξης και εξ αυτού γιατί και αν εξετάσουμε τις ε, παλιές χώρες μέλη, πάλι θα δείτε μια κατάσταση. Και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, επιδεινώνει την κατάσταση αυτή, η διαφοροποίηση δηλαδή. Γιατί δεν μπορεί να περιμένει κανένα να έχετε σε ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πολιτική της έκτη και σε ένα άλλο τμήμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν γίνεται αυτό γιατί αυτό συγχαίει την κατάσταση. Κατόπιν, η πηγή της κρίσης στις ε, χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι οι αγορές. Οι αγορές, με λίγες εξαιρέσεις. Και μια που η κρίση βασίζεται στην αγορά και τα μέσα αντιμετώπισης κρίσης θα πρέπει να βασίζονται στην ίδια αυτή την αγορά. Εκτός αυτού, βλέπουμε ξεκάθαρα και ανάφεραν κάποιοι εμπειρογνώμες αυτό, ότι όσο πιο καλύτερη ήταν η μακροοικονομική πολιτική πριν από την κρίση, τόσο καλύτερα οι χώρες αυτές μπορούσαν να αντέξουν τουλάχιστον το πρώτο στάδιο της κρίσης. Χαμηλότερα δηλαδή ελλείμματα δημοσιονομικά, να, μην υπάρχει δηλαδή χρέος κρατικό, να υπάρχει καλή εποπτεία της αγοράς, ε, ανακεφαλαιοποίηση κλπ. Τρίτον, ή ίσως δύο β' θέλετε. Έχουμε καταβάσει δύο συστήματα επιτηρήσει στα κράτη-μέλη, σταθερή ισοτιμίας κατά κάποιο τρόπο και ε, Point of view, Και κειμενόμενες ισοτιμίες. Τα σταθερά επιτόκια ε, οδηγούν σε καλύτερες μακροοικονομικές πολιτικές. Μπορούμε να δούμε χώρε που έχουν σταθερά επιτόκια χωρίς τα μέσα των, της διακοινόμενης να προχωρούν πολύ καλύτερα. Το τρίτο, κίνδυνοι και βλέπουμε διαφορετική αντίδραση στα κράτη, νέα κράτη-μέλη και διαφορετικές επιπτώσεις στα νέα κράτη-μέλη. Ο κοινός προγραμματής είναι το υψηλό επίπεδο κινδύνου και αυτό απορρέει από τις διαφορές των μακροοικονομικών παραμέτρων μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών. Πολύ λιγότερες δυνατότητες παρέμβασης, των προπολογισμό σε αυτή τη χώρα, μεγαλύτερη δυνατότητα περικοπής των δαπανών και είδαμε ότι σε πολλά από τα νέα κρατημέλη οι δαπάνες του προβλησμού είναι πιο ευέλικτες από ό,τι στα παλιά. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με το πάνελ όσον αφορά τις ε, αλλοδαπές ε, κεφαλαιοχικές επενδύσεις, ε, γιατί θεωρώ ότι αυτές ε, δεν είναι μια αηφόρα κατανάλωση. Ο πρώτος διακόπτη μπορεί να φτάσει σε μια ερώτηση. Uh, uh, Τέλος, σαν συμπέρασμα από την κρίση αυτή θα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι περισσότερες από τις νέες χώρες μέλη δεν έχουν τόσες ανάγκες για ε, βοήθεια στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών, εκτός από τις τρεις γνωστές χώρες, έχουν μάλλον ανάγκες για την ενίσχυση της οικονομίας, πλευράς αγοράς δηλαδή, από εκεί που προήλθαν τα προβλήματα. Και πάλι έχουμε το ευρώ, γιατί να, για να έχουμε ένα ενιαίο νομίσμα θα πρέπει να έχουμε οικονομική σύγκληση που δεν είναι. Αυτό που θα πρέπει να είναι είναι να υπάρχει μια διαφανής πολιτική στα κράτη-μέλη για να επενδύσουμε καλύτερα σε καλύτερες οικονομικές πολιτικές. Ευχαριστώ όλοι Σμιτ. Very Ευχαριστώ πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε στους, ε, ε, στα μέλη του πάνελ και να ακούσουμε και τη συζήτηση εδώ. Ποια προσθέμουν Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ελέγχθη ότι θα ήταν σταθεροποιητική η θέση εάν ε, περισσότερε χώρε μέλη θα μπορούσαν να έχουν εντεχθεί στο ευρώ πιο ομαλά. Δεν θέλω να μου το σχολιάσετε παρακαλώ. Ο κύριος Ντάρβας μάλιστα λέει στα συμπεράσματά του ότι η κρίση στην Ελλάδα ε, κατέστησε πιο δύσκολη την διεύρυνση της Ευρωζώνης. Γιατί Τον αντίον χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, εις βάθος συνεργασία στην Ευρώπη. Αν υπήρχαν λοιπόν κάποιες προτάσεις που να λένε ότι θα μπορούσαμε όχι να αλλάξουμε ριζικά, αλλά να διευκολύνουμε κάπως νέες χώρες να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Δεν πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγούσε σε γλίγορες αλλαγές. Γιατί το νέο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει νέες ε, νομισματικές πολιτικές Διαφυσβητούν ε, τις παλιές. Τα πράγματα κινούνται λοιπόν πολύ γλίγορα, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Μήπως είστε κάπως υπερβολικά απεσιόδοξος. Και μετά για αυτές τις διακοινωμενόμενες ισοτιμίες. Εγώ είμαι φιλελεύθερος και θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον να λέτε εσείς ότι αυτή η ελεύθερη ισοτιμία είναι προσθέμενη αξία. Εγώ νόμιζα ότι ακριβώς αυτό, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι ένας κακός τρόπος πολιτικών. Εγώ είμαι σε μια χώρα που εδώ και 40 χρόνια εξάγουμε τα προβλήματά μας υποτίμησης και λοιπά υπόλοιπη πόλη της Ευρώπης. Στους γειτονιούς μας κύριε, στη Δανία, στην Φιλανδία δεν είναι αλληλεγγύη αυτό. Δεν, κα... κατα... δεν οικοδομείται η Ευρώπη κατά αυτόν τον τρόπο έτσι. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Σπίν. 30 δευτερόλεπτα, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα Μα κοιτάξτε, αυτή η διακύμαση οδηγεί στις προνομιτικούς σταθεροποιητές στην οικονομία. Εγώ είπα ότι ακόμα και αν υπάρχει σταθερή ισοτιμία, παρά αυτά θα πρέπει να δούμε σε τι επίπεδο είναι. Ευχαριστώ πολύ. Οι εμπειρογνώμονες τώρα θα παρακαλώ να απαντήσουν. Δύο λεπτά ο καθένα γιατί έχουμε και ένα άλλο γύρο, ένα άλλο γύρο ερωτήσεων. Για να μπορέσει και η κυρία Μπερές και άλλοι. Κύριο Ζέλια παραδείγματο κάτι. Θα ακούσουμε τις απαντήσεις τώρα στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων και μετά θα περάσουμε στο τρίτο γύρο των ερωτήσεων. Προτιμάτε να συλλέξουμε όλες τις ερωτήσεις πρώτα ή να έχουμε ένα νέο γύρο. Okay. Όλες μαζί, εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι. Ε, θα ήθελα να ζητήσω, που δεν, συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ παρούσα από την αρχή, και θα επανέλθει σε τρία σημεία. Πρώτον, αν δεν εξετάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής καθεαυτής, αλλά ακούγοντας συζητήσεις που είχαμε και που έχουμε για την εισαγωγή ενός συστήματος εποπτείας των τομέων τραπεζών και ασφαλίσεων βλέπουμε πόσο η σημασία των τραπεζών αυτών και των ε, εξωτερικών κεφαλαίων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της συζήτησης. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε η κυρία Σμίτκοβα, ότι δεν ήταν τόσο ουσιαστικό στην κρίση. Εγώ έχω την εντύπωση να τον κοιτούμε την εκκίνηση της κρίσης στην Ουγγαρία, το γεγονός ότι συνέπεσε με την υιοθέτηση της υποστήριξης από τα κράτη-μέλη στον κραπεζικό τομέα είναι νομίζω ένα στοιχείο που πρέπει να λεφθεί υπόψη. Μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ένταξη των χωρών αυτών, ο μόνος περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων που αναφέρθηκε ήταν το θέμα κοινή των γεωλόγου που γνωρίζουμε πολύ καλά. Η ερώτηση μου είναι εξή. Δεν θέλω να μου δώσει αριθμητικά στοιχεία εδώ και τώρα, αλλά μεταξύ του δυσκόλου του ελέγχου και της εθνικής εποπτείας των αλλοδαπών τραπεζών και της πληθυκότητας των ε, δεσμευμένων κεφαλαίων τα πλεονεκτήματα ουσιαστικής επένδυσης των επιδείξεων αυτών ποιος είναι ο λογισμός δηλαδή, που έχετε δηλαδή από την άλλη μεριά πολλά κεφάλαια που μπαίνουν από την άλλη μεριά δεν ελέγχεται σωστά η αγορά αυτή, ποιος είναι ο τον στον οποίο καταλήγεται. Δεύτερον, για τις χώρες αυτές, και αυτό ισχύει και για χώρες της Ευρωζώνης, Έχουμε ένα πρόβλημα του μοντέλου που πρέπει να αναφερθεί και πολύ, το θέμα των ακινήτων στην Ιρλανδία και στην Ισπανία. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα προσαρμογής, γιατί ε, κάποια στιγμή η Ιρλανδία και η Ισπανία ήταν πρότυπα για επενδύσεις στην ε, περίοδο ανάπτυξης, το, δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Τώρα το πρόβλημα είναι που έρχονται τα πράγματα. Εσείς ε, πώς βλέπετε τα πράγματα στις χώρες της Βαλτικής όσον αφορά το μέσο όρο ανάπτυξης σε επόμενες Και τρίτη χώρα όσον αφορά την ένταξη ζώνη ευρώ. Και ζητώ συγγνώμη αν αυτό ελέγχθη ίσως στην αρχή. Εσείς πώ βλέπετε τα πράγματα σήμερα, γιατί πριν από την κρίση, ένα από τα στοιχεία ήταν ότι οι χώρε που βρίσκονται στην Ευρωζώνη δεν σέβονται τα κριτήρια. Γιατί να ζητάμε τώρα από μια νέα χώρα να τα σέβεται. Γιατί άμα δούμε τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μέλη, εσείς Πώς βλέπετε τον ορισμό των όρων διεύρυνσης της Ευρωζώνης και το συμφέρον των χωρών αυτών για την γλίγορη ένταξή του στην Ευρωζώνη. Ε, κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν και εγώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί ήρθα αργά και δεν άκουσα όλες τις παρουσιάσεις. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σχολιάσω. Fully said that, uh, Συμφωνώ, τελέχθη, ότι ε, οπωσδήποτε και οι κυβερνήσει πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του, ιδίω όσον αφορά την φορολογία. Εγώ είμαι από τη Λετωνία και ε, ευτυχώ τύχαμε τι αρρωγή για το ισοζύγιο πληρωμών. Δεν συμφωνώ όμω όσον αφορά το ότι οι χώρε τη Βαλτική δεν είχαν ισορροπημένη φορολογική πολιτική στη Λετωνία τονία υπήρχε στην, ε, δεν υπήρχε πάνω από το 30% το, ε, μέχρι το 2007 είχαμε πλεόνασμα στον προπολογισμό μας, πράγμα που δεν συμβαίνει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυρά δίνουν τόσα πολλά δάνεια που μέχρι το 2007 φτάσαμε στο 40%. Τώρα όμως λόγω της κρίσης με το ΕΠ φτάσαμε στο 200%. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί βέβαια θέμα της ισοτιμίας Αυτό που ενδιαφέρει κυρίω στις ε, σκαφιστικές ε, τράπεζες ήταν ένα τμήμα τη αγοράς. Εγώ ε, βλέπω ότι σε καλά χρόνια ορισμένε από τι σκανδιναβικέ χώρε είχαν 10% του χαρτοφυλακίου του στη Βαλτική με 30% κέρδου για όλο τον όμιλο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και όταν διαπραγματευθήκαμε την ε, συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με την Κομισιόν για την αργή στο ισοζύγιο ε, πληρωμών, ένας από τους όρους ήταν να κρατήσουμε τις τράπεζες αυτές και για το μέλλον, γιατί αν έχουμε πάνω από το 90% του εξωτερικού κεφαλαίου σε ευρώ, στη Λετωνία. Αν αυτό το χρήμα εξαφανιστεί δεν το ξαναβρούμε πουθενά. Είχαμε και την Paris Bank, BNB Paris. Και εγώ δεν αναφέρομαι εδώ στην ανάγκη περίσωση αυτής τη συγκεκριμένη τράπεζα, αλλά στην ανάγκη αποφυγή των στρεβλώσεων. Δηλαδή υπήρχε μια βοήθεια στην πλάτη των φορολογούμενων για τους επενδυτές στο εξωτερικό. Και γι' αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Κέλεμαν ότι ίσως θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε τη συμφωνία μας και να απομακρυνθούμε από την σταθερή ισοτομία, αν συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό. Και το δεύτερο θέμα αφορά την Εστονία. Κύριε Δάρας, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είχατε να πείτε και είδαμε κάποιες διαφάνειες πολύ ενδιαφέρουσες όσον αφορά την κατάσταση της Εστονίας και το ότι κανένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν τηρούν τα κριτήρια της Κοπεγάγης, αλλά η Εστονία θα το καταφέρει μάλλον φέτος. Και ο κύριος Επίτροπος Αλμούνια είχε πει ότι αν δεν γίνει τίποτα το τραγικό το μεταξύ, η Κομισιόν τον Ιούνιο θα καλέσει την Εστονία να ενταχθεί Εάν όμως η Εστονία τηρεί τα κριτήρια και δεν ε, τη δεχτείτε στην Ευρωζώνη, ποια είναι τα, τα μηνύματα που θα αποσταλούν. Θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωζώνη η Εστονία που είναι η μόνη χώρα που τηρεί τα κριτήρια του Μαστρέχη. τρέχει. Uh, uh, Μόνο τέσσερα λεπτά δίνω στον καθένα για τις απαντήσεις. Κύριε Ντάρβας, μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς. περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν τη διεύρυνση της Ευρωζώνης και κάποια συναφή θέματα. Ερωτήθηκε κατά πόσο το ελληνικό πρόβλημα, η κατάσταση στην Ελλάδα, διευκολύνει να δυσχεράνει τη διεύρυνση της Ευρωζώνης. Εγώ είμαι οικονομολόγος, όχι πολιτικός. Αν ήμουν πολιτικός όμως και είχα την ευκαιρία να διαθέσω χρήματα το φορολογουμένο για να σώσω μια χώρα και να μπορέσει να μπει στην ε, Ευρωζώνη και χρειάστηκε να δώσω ε, αναλυθεί απατηλά στοιχεία που να δίνουν καλύτερη δημοσιονομική εντύπωση χώρα, θα δίσταζα να το κάνω. Δεν είμαι πολιτικός, αλλά φοβάμαι ότι οι πολιτικοί των χωρών των, της ζώνης ευρώ ίσως πιστεύουν ότι αρκετά εσωτερικά προβλήματα έχουν και το να διευρύνουν την ευρωζώνη και να προσκαλέσουν νέα μέλη που έχουν σημαντικό χρέο. γιατί έχουμε και άλλε χώρε Ευρωζώνη με προβλήματα. Την Ισπανία, την Πορτογαλία. Για άλλου λόγου, όχι για του ίδιου λόγου ε, για τους οποίους η Ελλάδα αντιμετωπίζει κρίση που ήταν μια ανευθυνότητα δημοσιονομική. Η Πορτογαλία μπήκε το 1999 μετά από μια σημαντική περίοδο ανάπτυξης. Παρόμοια με αυτή που αντιμετωπίζουν οι Βαλτικέ χώρες ε, το τελευταίο καιρό. Υπήρξε υπερχρέωση, αλλά μεγάλη ανταγωνιστικότητα και μια οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια, όταν η Πορτογαλία μπήκε στο, στην Ευρωζώνη, είχε το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Τώρα, η Ισπανία εξαιτία τη μείωση των επιδοκίων και κάποια θέματα χώρε πολιτική ε, παρουσίασε μια τεράστια άνθηση στη στέγαση, τεράστια αύξηση την κατανάλωση και διόγκωση του κατασκευαστικού κλάδου. Μεγαλύτερη ανάπτυξη του, στεγαστικού, του κατασκευαστικού κλάδου στην Ισπανία από οπουδήποτε αλλού, αλλά παρόλα αυτά και η Ισπανία αντιμετωπίζει προβλήματα και δύσκολα θα ξεφύγει από την κρίση. Γιατί στο μεταξύ έχασε και ένα τμήμα τη ανταγωνιστικότητά και σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους ε, υπήρχε πρόβλημα. Η Πορτογαλία μπήκε μετά το 99 βέβαια, αλλά εξαιτία της διάστασης, των διαστάσεών της αντιμετωπίζει μικρότερα προβλήματα από την Ισπανία. Οπότε πολύ πιο διστακτικά οι χώρες Ευρωζώνης θα επιτρέψουν διεύρυνση για άλλες χώρες που ίσως επίσης δημιουργήσουν προβλήματα αργότερα. Από πολιτική άποψη ήμουν και εγώ πιο αυστηρός με τις νέες χώρες δεδομένων των προβλημάτων που είχαμε στο παρελθόν. Δεν ξέρω ποιος είπε προηγουμένως, ο κύριος Κέρεμας, ότι στις νέες χώρες η αγορά εργασία και προϊόντων είναι πιο ελαστικές από ό,τι στις παλιές χώρες. Οπότε αυτήν την άποψη υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες διεύρυνση, αλλά και είναι επικίνδυνη μια τέτοια διεύρυνση ευρωζώνης. Τώρα, για το κατά πόσο η Πολωνία έχει συμφέρον να κρατήσει κειμενόμενε ισοτιμίε. Το θέμα είναι ότι η Πολωνία έχει αποκτήσει μεγάλη αξιοπιστία λόγω των καλών τη επιδόσεων και έχει και πολλά λαμπρό μέλλον. Τώρα για τι βαλτικέ χώρε, νομίζω ότι συμφέρον του είναι να μπουν στην Ευρωζώνη το συντομότερο δυνατόν. Το θέμα τη ανταγωνιστικότητα όμω για αυτέ είναι πολύ σοβαρό. Φοβούμαι ότι θα μπουν και αν η Εστονία μπει με, με την ισχύουσα ισοτιμία θα γίνει μια δεύτερη Πορτογαλία. Είναι ελαστική η Εσθονία, αλλά αν δείτε την πτώση, την ονομαστική μείωση των μισθών, ιδιαίτερα τελευταία οκταετία, είναι πολύ μικρό το ποσοστό στην Εστονία. Γιατί μειώσει μισθών υπάρχουν παντού, αλλά στην Εστονία είναι σχετικά μικρό το ποσοστό. Δεν νομίζω ότι όμω ότι με αυτό το μέτρο, με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τη Εστονία. Και αν μπει στην Ευρωζώνη θα μπει ε, με, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο. Βέβαια είναι μικρή χώρα. Πάντως το θέμα της ανταγωνιστικότητας είναι το πιο σοβαρό για τη χώρα αυτή και θα πρέπει να το εξετάσει. Στο πάνελ συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχουν δύο είδη μοντέλων ανάπτυξης. Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη είχαμε οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη αύξηση της ανταγωνιστικότητας του μεταπητικού κλάδου και αύξηση των εξαγωγών. Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, ένα μεγάλο τμήμα των κεφαλαίων απορροφήθηκε από το στεγαστικό κλάδο και εκεί υπήρξε ένα boom στα ακίνητα, κάτι που δεν βοήθησε οι να ξεφύγουν από την κρίση. Υπάρχει διαφορά στο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της κεντρικής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Χρειάζεται μια μικρή αλλαγή, αλλά όχι μια ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση. Ο κύριος Κέρεμαν, σε ευχαριστώ. Υπήρξε ερώτηση της κυρίας Γιακονσάρη για τις πολιτικές διαστάσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν καλύτερα την κρίση. Μπορεί να σα απογοητεύσω, αλλά δεν θα επιμείνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν μελέτε που εξετάζουν τι είδου ε, συνασπισμού ή ενιαίου κόμματο ε, είναι καλύτερε για τι πολιτικέ και ποιε επιπτώσει έχουν τα μέτρα του στην οικονομία και στην ε, οικονομική ανάπτυξη. Δεν πρόκειται να το αναλύσω εγώ αυτό γιατί υπάρχουν έγκυρες επιστημονικές μελέτες για τέτοια θέματα. Εσείς αναφέρετε στην Πολωνία και είπατε πώς μπορούμε να διδαχθούμε από, τις, ε, από τη σωστή αντιμετώπιση της κρίσης από τη χώρα αυτή. Θα πρέπει να δούμε καταρχήν τα χαρακτηριστικά αυτής της χώρας. Αναφέρθηκε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό ήταν μια υγιής δημοσιονομική πολιτική. Η Πολωνία είναι σχετικά μεγάλη χώρα και σχετικά κλειστή οικονομία. Μόνο το 40% του εμπορίου μόνο το, μόνο το εμπόριο αντιστοιχεί μόνο σε 40% του εμπορίου. Σε σχέση με άλλες χώρες είναι μικρό το ποσοστό. Επίσης δεν υπήρξαν τόσο μαζικές επενδύσεις σε τοξικά ε, προϊόντα, γιατί ήταν αρκετά συντηρητικό το τραπεζικό σύστημα. Βέβαια το ότι μια οικονομία είναι μεγάλη και σχετικά κλειστή δεν σημαίνει ότι βρίσκεται κανείς στο απειρόβλητο της κρίσης. Παράδειγμα η Ρουμανία. Σχετικά μεγάλη χώρα, όχι σε την Πολωνία βέβαια. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν το άνοιγμα στο εμπόριο. Παρόμοιο άνοιγμα στο εμπόριο με την Πολωνία και παρόλα αυτά η Ρουμανία επλήγει από την κρίση πολύ σοβαρότερα από την Πολωνία. Ο κύριος Ζήλε ρώτησε ίσως θα πρέπει να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση της κλειδωμένης ισοτιμίας της Λετωνίας. Αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, αν χρειάζεται τέτοια αναδιαπραγμάτευση, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά στοιχεία. Μια υποτίμηση ίσως ήταν καλή, μια υποτίμηση του νομίσματος, γιατί θα αυξηθούν οι εξαγωγές. Και ένα από τα προβλήματα της Λετωνίας ήταν το τεράστιο έλλειμμα που είχε στο ισοζύγιο. Γιατί είχε πολύ περισσότερε εισαγωγέ από ό,τι εξαγωγέ. Χρειάζεται να αυξήσει τι εξαγωγέ για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέο τη. Οπότε μια υποτίμηση του λετωνικονομίσματο θα ήταν καλό από την άψη γιατί θα αναζωογονούσε τι εξαγωγέ. Υπάρχει όμω και το θέμα της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών οι υποθήκες ή τα δάνεια των επιχειρήσεων είναι σε ευρώ, οπότε η αποπληρωμή θα είναι πολύ πιο ακριβή αν γίνει υποτίμηση. Θα αυξηθεί κατά 30-40% το χρέος που είναι εκφρασμένο σε ευρώ. Οπότε αυτήν την άποψη αντεδείκνυται μια υποτίμηση. Επίσης το κλείδωμα της ισοτιμίας με το ευρώ ίσως δεν είναι και τόσο καλό για το λετωνικό νόμισμα. Ίσως δώσει το μήνυμα ότι η πολιτική σταθεροποίηση της ισοτιμίας και η προετοιμασία για την εισαγωγή στο ευρώ δεν είναι και πολύ δόκιμη λύση. Και πάλι μου επισημαίνουν ότι εξάντλησα το χρόνο μου. Λένε ότι να μην ασκήσει, να διαρκέσει μια διετία το ΑΕΡΕΜ, να πάει κατευθείαν σε κλείδωμα της ισοτιμίας. Πάντως δεν υιοθετήθηκε αυτή η πολιτική. Πρέπει να ολοκληρώσω. Ναι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και την κυρία Σμίτκοβα. Ευχαριστώ. Τρία σχόλια. Το πρώτο αφορά το ρόλο της εποπτείας. Έγινε πολλά σχόλια στη συζήτηση για το θέμα αυτό και μέχρι στιγμής δεν αποδώσαμε τη δέουσα προσοχή στο ρόλο της εθνικής εποπτείας στη διάρκεια της κρίσης. Βέβαια, οι αλλοδαπέ Τράπεζε ε, βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν και τον κίνδυνο. Οπότε η Εθνική Εποπτική Αρχή έχει ω ρόλο τον περιορισμό του κινδύνου. Ο υπόπτη θα πρέπει να εντοπίσει τους συστημικούς κινδύνους και τους μακροοικονομικούς κινδύνους μια χώρας και να διαπραγματεύσει προστατευτεί με τις αλλοδαπές τράπεζες, οπότε να γίνει ένα είδο εσωτερήκευσης του κινδύνου στο σύστημα διαχείρισής τους. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η ανάμειξη των αλλοδαπών τραπεζών αυξάνει το κίνδυνο έκθεση στη, στις του συναλλάγματος. Αλλά είναι ρόλο τη Εθνική Αποπτική Αρχή να κάνει σωστέ διαπραγματεύσει με τι ε, αλλοδαπέ τράπεζε. Σε ό,τι αφορά τι Βαλτικέ χώρες ήταν υγιεί και υπεύθυνε οι δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά ο ιδιωτικό κλάδος ήταν αυτό που έδειξε ανευθυνότητα. Αλλά και εκεί θα πρέπει η αποπτική αρχή να μην αφήσει τις τράπεζες να υπερεκτεθούν σε τέτοιους μακροκινδύνους. Γιατί ήταν υπερχρεωμένος ο ιδιωτικός κλάδος Εκεί έπρεπε να είναι πιο αυστηρέ οι εποπτικέ αρχέ τη διαπραγματεύση του με, με το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αλλιώ πώ θα έχουμε έναν υπεύθυνο δημόσιο κλάδο, αν ο χρηματιστικό τομέα ε, ενισχύει την τάση του ιδιωτικού κεφαλαίου να υπερχρεώνεται. Άλλο πρόβλημα ήταν η απειρία των νοικοκυριών στις νέε χώρες μέλη, γιατί δεν έχουν καλή οικονομική παιδεία τα νοικοκυριά στι νέε χώρε. Στην ε, Εθνική Τράπεζα τη Τσεχία είχαμε εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα ε, της εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα τα νοικοκυριά και να αποφευθεί η υποχρέωσή τους ε, και η έκθεση τους στο μέλλον. Εξαρτάται και από το κράτος ε, πώς θα βελτιώσει την ενημέρωση και την διαπαιδαγώγηση του κόσμου ώστε να αποφευθεί ο κίνδυνος. Υπάρχει και διαφορετική νοοτροπία και πολλές διαφορές. Δεν είμαι εμπειρογνώμονα σε θέματα πολιτικής οικονομίας, πάντως ο ρόλος των θεσμικών οργάνων στις χώρες αυτές δεν είναι ο ίδιος. Στις νέες χώρες μέλη η κεντρική τράπεζα είναι ανεξάρτητη. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τα θεσμικά όργανα όπως ε, από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Επιβεβαιώθηκε η ανεξαρτησία της Εθνικής Τράπεζας στις νέες χώρες. Οπότε σε αυτές τις χώρες η νομισματική πολιτική είναι και πιο αξιόπιστη. Οπότε σίγουρα τα θεσμικά όργανα δραματίζουν ρόλο για την ε, αύξηση της αξιοπιστίας. Τώρα, κατά πόσο ε, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και κειμενόμενη ισοτιμία. Και πάλι εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά μιας χώρας. Αν πρόκειται για μια συγκλίνουσα οικονομία, που δεν έχει πολύ ελαστική αγορά εργασίας και αν άλλε ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ανοιχτέ ε, αγορές εργασίας προς τη χώρα αυτή, τότε μια κειμενόμενη ισοτιμία αντισταθμίζει κάπως μια ανελαστική αγορά εργασίας και βοηθά τη χώρα και στη διαδικασία σύγκλησης αλλά και στην ε, αντιμετώπιση των κινδύνων, των κλειδονισμών. Αν εμείς οικονομία και δεν μιλάω για ανταγωνιστική υποτίμηση, αλλά αν υπάρχει ένα ελαστικό σύστημα που επιτρέπει σε μια οικονομία νέα χώρα να συγκλίνει καλύτερα, ίσω μια κειμενόμενη ισοτιμία δεν θα ήταν κακή ιδέα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του καλεσμένου μα για τις ε, πολύ αξιόλογες ομιλίες τους στα πλαίσια του πρώτου πάνελ και να περάσουμε στο δεύτερο με τους καλεσμένους μας ε, εμπειρογνώμονες Χάιλ και Ζουλέγκ. Το δεύτερο πάνελ αφορά τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στη στρατηγική εξόδο από την κρίση. Ο εμπειρογνώμονα μας είναι ο κύριος Πίτερ Χάιλ από το γραφείο του Πρωθυπουργού, τέο υποδιευθυντή του Εθνικού Οργανισμού Ανάπτυξης της Ουγγαρίας και ο κύριος Φάμπιαν Ζουλέγκ, αναλυτής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτική. Θα εφαρμόσουμε του ίδιου κανόνε με το προηγούμενο πάνελ. Έχετε 10 λεπτά για την κάθε παρουσίαση και θα ακολουθήσει γύρω σε ερωταπαντήσεων. Κύριε Χάιλ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ε, προέρχομαι από ένα ε, κρατικό οργανισμό, θα σας μιλήσω ως εμπειρογνώμων, για τον ρόλο της πολιτικής συνοχής μετά την κρίση. Κάτι που είναι επίκαιρο. Οι ερωτήσει που μα τέθηκαν πριν από την έρεξη του σεμιναριού είναι κατά πόσο η πολιτική συνοχής μπορεί ή ε, μπορεί να είναι ή υπήρξε βασικό ε, στοιχείο για την αντιμετώπιση της κρίσης από τις χώρες μέλη. Ποιος ήταν ο ρόλος της στις νέες χώρες μέλη και πώς μπορεί μακροπρόθεσμα η πολιτική συνοχή να ε, συνδεθεί με μια στρατηγική εξόδου από την κρίση, αλλά και τι ρόλο θα παίξει για το 2020. Τα θέματα εν προκειμένου είναι πρώτα ποια ήταν η επίπτωση της κρίσης από την πλευρά της πολιτικής συνοχής, ποια ήταν η ανταπόκριση της πολιτικής συνοχής και στο επίπεδο της Ένωσης αλλά και των χωρών μελών και δοθήσεις της καταστάσεως όπου βρισκόμαστε αλλά και της ε, συζήτηση που αρχίζει για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική. Ε, χρειαζόμαστε διαφορετική πολιτική ή η πολιτική συνοχή μπορεί να εξυπηρετήσει και για το μέλλον. Το συμπέρασμά μου θα είναι, από τώρα σας το λέω, το συμπέρασμά μου θα είναι ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Μπορεί να προσαρμοστεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε Πρώτα λοιπόν ποια υπήρξε η επίπτωση της κρίσης, ποιες ήταν οι προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε. Έχει βελτιωθεί βέβαια κάπως η κατάσταση, αλλά ο βασικός ρόλος της συνοχής είναι να μειώσει τις αποκλήσεις μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Η επίπτωση ήταν διαφορετική δεν ξέρω, δεν θέλω τώρα να κάνω ε, διακρίσεις μεταξύ παλαιών και νέων χωρών μελών και διάφορες κατηγορίες που υπάρχουν, αλλά είναι σημαντικό αν εξετάσει κανείς την μελέτη της Επιτροπής που έχει γίνει για τις περιφέρειες για το 2020, θα δείτε και πιο μακροπρόθεσμα τις νέες προκλήσεις που είναι για παράδειγμα κλιματική αλλαγή, ε, ασφάλεια της ενέργειας, διατήρηση των κοινωνικών συστημάτων. Θα δείτε ότι όλα αυτά έχουν διαφορετικές επιπτώσεις αναπεριφέρεια στην Ένωση. Και μέσα στην ίδια την ε, κρίση είχαμε ε, διαφορετικά σοκ. Όλες οι χώρες αντιμετώπισαν ε, την μείωση της πίστης, την μείωση της απασχόλησης. Πολλές χώρες μέλη αντιμετώπισαν και προβλήματα με τα ισοζυγιά τους. Στις νέες χώρες μέλη, επειδή είναι χαμηλότερα στην οικονομική ανάπτυξη, σε πολλές περιπτώσεις ήταν λιγότερο ανταγωνιστικές, οι υποδομές τους είναι λιγότερο, αλλά και οι διαθρώσεις τους είναι λιγότερο ενισχυμένες και είχαν και σε περιπτώσεις, σε περιπτώσεις και προβλήματα ε, ασφάλειας της προμήθειας της ενέργειας. Μιλήσαμε συχνά για την Ουγγαρία όπου είχαμε υψηλό επίπεδο ε, κρατικού χρέους, μειωμένη πρόσβαση στο διεθνές κεφάλαιο στα πλαίσια της ε, κρίσης. Για πολλά χρόνια γίνονται προσπάθειες δημοσιονομικών διορθώσεων με πακέτα λιτότητας το ένα μετά το άλλο, που έχουν ωστόσο μειώσει την δυνατότητα κινήσεων της κυβέρνησης ό,τι αφορά τις πολιτικές δαπανών και βέβαια και χαμηλή απασχόληση. Πώς μπορεί τώρα η πολιτική συνοχή να απαντήσει σε τέτοιες περιπτώσεις και από την πλευρά της Ένωσης αλλά και από την πλευρά των χωρών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε ένα πακέτο για την αντιμετώπιση της κρίσης στα τέλη του 2008 που πολλά μέτρα τα οποία ήταν ειδικά κομμένα και ραμμένα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση από πλευρά πολιτική συνοχή. Η Κομισιόν προσπάθησε πρώτα να κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα ταμεία τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από πλευρά κυβερνήσεων για παρέμβαση που αυτά έλεγε τότε η ε, κοινή γνώση, εν πάση περιπτώσει, για το πώ πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση. Οι προκαταβολέ που έγιναν από τον κοινοτικό προπολογισμό στι χώρε μέλη αυξήθηκαν. Η Κομισιόν ε, πρόσφερε τη δυνατότητα να γίνει το λεγόμενο front loading στη διάρκεια αυτή με, από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Παρατάθηκε και η διάρκεια προγραμμάτων με ε, τον, που είχαν τον κίνδυνο βέβαια να χάσουν ε, κονδύλια λόγω της κρίσης και υπήρξαν και πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πήραν τη μορφή νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ενισχύσει τα μέτρα αυτά. Δεύτερο, πρόσφερε η Κομισιόν τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να αλλάξουν προγράμματα που μόλις είχαν εγκριθεί, αλλά βέβαια άλλαξαν τα βασικά στοιχεία στα οποία βασίζονταν. Και αυτό έδειξε μια ευκαμψία και μια προσαρμοστικότητα από πλευρά ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δηλαδή τα προγράμματα έπρεπε να αλλάξουν, μπορούσαν να αλλάξουν. Υπήρξε και μια ανταπόκριση για να αλλάξει το ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής. Κάτι το οποίο ίσως είναι ασυνήθιστο μόλις το δεύτερο έτος της εφαρμογής του, πλαισίου, του δημοσιονομικού πλαισίου. Πολλά μέτρα υιοθετήθηκαν που υποτίθεται ότι θα διευκόλυναν την κατάσταση των απολυπτών. Δεν θα τα πω όλα τα μέτρα αυτά, αλλά είχαν μετρήσιμη συγκεκριμένη ε, επίπτωση στους απορρίπτε, beneficiaries. Έγιναν και ορισμένα, υπήρξαν και ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Ένα θέμα που θα έπρεπε να τονιστεί εδώ νομίζω έχουμε κάποια πράγματα που δεν σκεφτήκαμε σχετικά με το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει το Ταμείο Συνοχής ως όργανο ανάπτυξης. Θα έπρεπε να γίνει πιο εύκαμπτο και να επιτρέπεται να χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, και μέτρα βελτίωση τη αποδοτικότητα τη ενέργεια, κάτι το οποίο επί του παρόντο δεν είναι δυνατόν. Οι χώρε μέλη ανταποκρίθηκαν με διαφόρου τρόπου. Έχουμε στατιστικέ βασισμένε σε μια δημοσκόπηση ε, με συνεργασία συναδέλφων από άλλε χώρε μέλη. 11 τουλάχιστον χώρε μέλη άραξαν τα προγράμματά του σε κάποιο βαθμό. Όπω για παράδειγμα στην Ουγγαρία προσπάθησαν να πάρουν χρηματοδότηση και να την δώσουν σε μικρές και μεσές επιχειρήσεις από αλλού σε μια προσπάθεια να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα, την ε, θέση των απολυπτών, των δανείων και στην περίπτωση της Ουγγαρίας δόθηκαν και αποζημιώσεις για τις αλλαγές της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Και επίσης ε, για, έγινε μια προσπάθεια για την μείωση ή για την αποζημίωση, αν θέλετε, λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων. Θα μπορούσαμε εν όλο να πούμε ότι η γενική ανταπόκριση στην κρίση ήταν αύξηση των κρατικών δαπανών και εκεί έπαιξε ένα ρόλο το Ταμείο Συνοχή, χρησιμοποιώντα κάθε δυνατότητα που υπήρχε για να αυξηθεί η ρευστότητα στι αγορέ και ιδιαίτερα στι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Όπου αυτό ήταν αναγκαίο, επαναπρογραμματίστηκαν τα ταμεία για να προσφερθούν περισσότερε δυνατότητε στον τομέα των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Όλα αυτά απαιτέλεσαν πραγματικά το κλειδί για χώρε όπω η Ουγγαρία, όπου χωρί χρηματοδότηση κοινοτική ο δημόσιο τομέα δεν θα μπορούσε να είχε ενισχύσει του οικονομικού φορεί. Υπήρξε σωστή, καλή συμβίωση λοιπόν ε, μεταξύ ε, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σκέψεων. Αυτά τι σημαίνουν τώρα για, το, για την πολιτική συνοχή και μέσα στα πλαίσια τη αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Παραδοσιακά η πολιτική συνοχή θεωρείται σαν ένα μηχανισμό αλληλεγγύη, αλλά έχει συνδεθεί με την Λισαβόνα ήδη για την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο, δημοσιονομική περίοδο και όσοι εργάζονται επί τόπου γνωρίζουν ότι με κανένα τρόπο δεν αποτελεί μηχανισμό για την αποζημίωση των φτωχών χωρών που ανοίγουν τις αγορές τους, που ανοίγουν τις οικονομίες τους αγορές η πολιτική συνοχή έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να αποβεί προ όφελο ολόκληρη της Ευρώπης. Η κρίση έδειξε καθαρά ότι η πολιτική συνοχή επίσης έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και βραχυπρόθεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι έχει διαφορετικές επιπτώσεις περιφερειακά. Είναι διαφοροποιημένε οι ανταποκρίσει σε διαφοροποιημένε προκλήσει. Εάν εξετάσει κανείς προς τα που κινείται η παρούσα συζήτηση σε σχέση με την Ευρώπη του 2020 αλλά και την αναθεώρηση του προπολογισμού, θα δείτε ότι η πολιτική του 2020 στην αρχική της μορφή δεν μιλούσε αρχικά για πολιτική συνοχή, σχεδόν καθόλου. Το Budget Review Paper, το οποίο αποσύρθηκε ευτυχώ, μείωνε την πολιτική αυτή σε σημαντικούς τομείς. Η εξήγηση είναι απλή. Η πολιτική συνοχής είναι και το δεύτερο μεγαλύτερο σημείο που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος λοιπόν θέλει μείωση τέτοιων χρηματοδοτήσεων πρέπει να στραφεί κατά της πολιτικής συνοχής. Αλλά οι προτάσεις που ακούγονται για την ώρα κινούνται προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός λένε ότι δεν είναι καλή ιδέα να γίνει προσπάθεια να καθιερωθούν νέοι μηχανισμοί ε, δαπανών εκτός της πολιτικής συνοχής Νομίζω εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει αποδοτικές πολιτικές δημοσίων δαπανών πρέπει να ρίξει ιδιαίτερο βάρος στην πολιτική συνοχή και να μην θεσπίσει νέους μηχανισμούς παρά όπου είναι απολύτως απαραίτητο. Για παράδειγμα, για την προστασία περιβάλλοντος ή για τις μεταφορές η ε, Ένωση δεν έχει πολιτικές, θεσμικές και κανόνες ούτε πρακτική εμπειρία ε, δαπάνης μεγάλων ποσών υπέρ τη οικονομία. Η μόνη πολιτική που μπορεί να το πράξει αυτό, που να το εξασφαλίσει αυτό για την ώρα, είναι η πολιτική συνοχή, διότι έχει στρατηγικό προγραμματισμό, διότι συγχρηματοδοτείται από τι χώρε μέλη και γιατί είναι βασισμένη και στην συνεργασία των, των, των ιδιωτικού και δημοσίου, αλλά και τη επικουρικότητας. Όλα αυτά δείχνουν ότι κινούμαστε προ ένα συμπέρασμα. Εγώ θεωρώ ότι η κρίση κατέδειξε ότι η Ευρώπη στο σύνολό της χρειάζεται μια πολιτική δημοσίων ταπανών. Η πραγματική ερώτηση είναι όχι τόσο αν μας αρέσει η Λισαβόνα ή όχι, αν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ε, αύξηση της ανεργίας ή όχι, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Για αν μας αρέσει η έρευνα και η ανάπτυξη, ο τρόπος είναι πώς θα εξασφαλίζουμε αυτά. Και νομίζω ότι, ο τρόπος, ότι η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε μια περίπλοκη ε, ε, πολιτική ανταπόκριση που θα έχει τη δυνατότητα να διοχετεύει μεγάλα ποσά χρημάτων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει και την απαραίτητη ευκαμψία ε, βραχυπρόθεσμα. Και αυτή θα είναι η πολιτική συνοχή. Χωρί να λησμονούμε και το πρόβλημα τη αλληλεγγύη. Νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτική συνοχή, να την επανακαθιερώσουμε ω ένα νέο είδο μηχανισμού και ίσω και να την ενισχύσουμε ω ένα πυλώνα τη οικονομική πολιτική. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάιλ. Κύριε Ζούλεγκ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα μια εισαγωγή εδώ με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής. Είμαστε ένα ανεξάρτητο think tank που βρισκόμαστε στην στις Βρυξέλλες. Μπορούμε να είμαστε δηλαδή επικριτικοί για κάποια θέματα. Δύο κύρια θέματα για το ε, ε, απόγευμα σήμερα. Αυτό που συγκύρωσε είναι η απόδοση μέχρι στιγμής ε, του μέσου συνοχή ε, σε σχέση με την ε, κρίση. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά εγώ θα πρέπει, θέλω κυρίως να δω προ τα που θα πάμε και τι θα κάνουμε προσεχώ. το μέλλον δηλαδή. Εντάξει, το κυρίε τις κύριες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις νέες χώρες, αλλά και στις παλιές χώρες μέλη. Πολλέ προκλήσει βράχη, μέσο και πρόθεσμα. Ακούσα ορισμένε. Έχω εδώ προετοιμάσει ένα κατάλογο όχι εξαντλητικό, αλλά υπάρχει για να βασίσουμε κάποια πολιτική. Ορισμένε είναι άμεση επίπτωση κρίση. οι περισσότερε όμως ε, χρονολογούνται από πριν από την κρίση. Μπορεί η κρίση να τι επιδίνωσε. υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών, τα ακούσαμε αυτά, αλλά είναι νομίζω σαφέ ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολο περιβάλλον για να προχωρήσουμε. Θα επανέλθω. Είναι τα κατάλληλα μέσα, τα μέσα αυτά συνοχή για να αντιμετωπίσουμε αυτού του τύπου τις προκλήσεις. Υπήρχαν ορισμένες αμφιβολίες ε, στο παρελθόν για την αποτελεσματικότητα των μέσων αυτών συνοχής. Βέβαια δεν έχουμε και πολλά άλλα στα χέρια μας για τα νέα κρατημέλη ιδίως. Μέχρι στιγμής ε, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι βοήθησαν τα μέσα αυτά ε, για την αντιμετώπιση της ε, κρίσης. Υπήρχε μια έρευνα της Επιτροπής των Περιφερειών που λέει ότι 55% των περιφερειών θεωρούν ότι οι επιπτώσεις είναι σημαντικές ή σχετικά σημαντικές. Για να δούμε για το μέλλον όμως, όσον αφορά τις ε, μελλοντικές κύριες προκλήσεις, υπάρχουν πέντε όροι νομίζω πρέπει να πληρούνται για να είμαστε σίγουροι ότι τα μέσα συνοχή ε, μπορούν να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Η κλίμακα της ε, ανταπόκρισης, ταχύτητα, δομή και ευελιξία για να μπορούν να αντιμετωπίσουν στις προκλήσεις πρέπει να υπάρχει προσθετικότητα, να υπάρχει συνοχή και αποτελεσματικότητα, ιδίως σε σχέση με άλλες πολιτικές και θα πρέπει να υπάρχει το σωστό παράθυρο ευκαιρίας. Θα επανέλθω σε αυτό. Καταρχήν, η διάσταση. Τα μέσα συνοχής είναι ένα μικρό τμήμα των δημοσίων δαπανών, 0,4% του ευρωπαϊκού ε, ΑΕΠ. Αλλά είναι, δεν είναι αλλά είναι πιο σημαντικά στις νέες χώρες μέλη, γιατί έχουν χαμηλά επίπεδα. Επίσης είναι πιο σημαντικό όταν εξετάζουμε τις ε, δημόσιες επενδύσεις και όχι τις ε, δημόσιες δαπάνες. Οι επενδύσεις είναι όσον αφορά, δηλαδή η παρεμβάση είναι όσον αφορά τις επενδύσεις ιδίως. Είναι ένα δώρο κατά κάποιο τρόπο γιατί δεν χρειάζεται να ε, ανταποκρίνονται στα έσοδα, δεν υπάρχει τόσο προστρέβλωση και υπάρχουν επιπτώσεις και στις δημόσιες και εν μέρει στις ιδιωτικές δαπάνες. Υπάρχει το από αυτό που αποκαλούμε front-loading στη σημερινή κρίση, ε, βραχυπρόθεσμα δηλαδή επειδή αλλά εξ αυτού και λιγότερα πόροι για το μέλλον. Και επίσης, συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, παιδί στην έρβα και την κρατομία επίσης στις Λοιπόν, η σημαντική η κλίμακα, αλλά εάν ε, δεν τις χρησιμοποιήσουμε παρκώς, δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις και από μόνοι τους δεν αρκούν. Τώρα, ταχύτητα, δομή και ευελιξία. Έγιναν διάφορες βελτιώσεις του συστήματος ε, για να αντιποκριθούν στην κρίση. Παρά αυτά θεωρώ ότι παραμένουν πολύ αργά και πολύ γραφειοκρατικά αυτά τα μέσα. Αυτό δεν αφορά μόνο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ορισμένε χώρε τα συστήματα είναι πιο δύσκολα από τι άλλε. Αυτό σημαίνει ότι γενικά δεν είναι πολύ εύκολα να μεταφερθούν τα χρήματα μεταξύ των προτεραιοτήτων και να προσθέσουμε νέε προτεραιότητε υπήρχε δυνατότητα αναθεώρηση των προγραμμάτων λόγω της κρίσης, αλλά και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί σε πολλές χώρες έχουν εμπλακεί πολλούς από τους ενδιαφερόμενους και αυτό είναι χρονοφόρο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει νέα κατανομή γεωγραφικά, δηλαδή χωρών ή περιφερειών οι δαπάνες ε, προσανατολίζονται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές, άρα μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι τρέχουσες επενδύσεις. Και έχουμε τον πολιετή χαρακτήρα επίσης. 2007-2013 είναι η προγραμματική περίοδος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν περισσότερη ευελιξία μετά το 2013. Αλλά όσον αφορά τις άμεσες επιπτώσεις της κρίσης θα είναι πολύ αργά για μετά το 2014 προσθετικότητα. οι δράσει του τομείου αυτού είναι συμπραγματικέ, δηλαδή οι δράσει που δεν θα λάμβανουν χώρα διαφορετικά. Μάλλον, γιατί υπάρχει έλλειψη ε, κρατικής ε, επένδυσης και υπάρχουν υψηλότερες ανάγκες. Ε, Υπάρχει επίσης μια τάση να υπάρχει μια κίνηση πιο πολύ στο mainstream, δηλαδή η χρηματοδότηση πιο βασικών προγραμμάτων. Στο παρελθόν ε, τα ταμεία αυτά χρησιμοποιούσαν για την επένδυση καινοτομικών προγραμμάτων, προγραμμάτων δηλαδή που θα, είναι, θα είχαν κατά τα άλλα ε, χρηματοδοτηθεί. Τώρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση που στηρίζει πιο βασικά προγράμματα. Και χρειαζόμαστε σε λιγότερο παραδοσιακές ε, περιοχές. Ε, παραδείγματος χάρη είναι ανάγκες για πιστώσεις, ε, επενδύσεις, επιχειρήσεις που δεν μπορούν να βρουν χρήματα από άλλο. συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Οι γενικές πολιτικές δηλαδή θα πρέπει να χρηματοδοτεί το μέσο συνεχής. Έχουμε το Ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης, υποστηρίζει εταιρείε, υποστηρίζει την αγορά εργασία, αυξάνει την ε, ζήτηση και επενδύσει στις υποδομές και όπως ελέγχθη ήδη, τα μέσα συνοχής εργάστηκαν πάρα πολύ καλά εδώ, πιο αποτελεσματικά ίσως όσον αφορά κυρίως τη μακροπρόθεσμα, δηλαδή αγορά απασχόλησης και ε, υποδομές και κάποιες πτυχές ε, της υποστηρίξης ε, των επιχειρήσεων. Ε, στα πλαίσια αυτά η μετατροπή σε μια ευφυή πράσινη συμπραγματική οικονομία, αυτό που λέγαμε τώρα Ευρώπη 2020, τώρα βλέπουμε εδώ στο μέλλον η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι πολύ σημαντική, θα επανέλθω σε αυτή. Επίση, η χρηματοδότηση μπορεί να ενδυναμώσει τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει ή τουλάχιστον να μην είναι σε αντίφαση με αυτέ. Ένα παράδειγμα, όταν κοιτάμε τι αγορέ εργασία, αν η χρηματοδότηση χρησιμοποιεί για να μειωθεί η προσφορά εργαζομένων, αυτό ίσως μεσο... Ε, βραχυπρόθεσμα βοηθήσει, αλλά όχι ε, μακροπρόθεσμα. Ε, βλέπουμε να επιταχύνεται η, δαπα, η, η εκταμιευσή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά ε, δαπανούνται σωστά. Το ένα δεν συνεπάγεται αυτόματα το άλλο. Παράθερο ευκαιρία. Ευρωπαϊκό Ταμείο Οικονομικής ε, Ανάπτυξης έδωσε κάποια κίνητρα, ιδίω φορολογικά, που θα πρέπει να είναι προσωρινά. Περισσότερες χώρες λένε ότι θα αποσυρθούν αυτά τα κίνητρα μετά το 2010. Και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουν τα χρήματα των ε, μέσων συνοχής να ξεκινήσουν να χορηγούνται. Το θέμα είναι ότι αν αρχίσουμε αυτή τη στιγμή θα περάσουν μήνες, αν όχι ολόκληρο χρόνο για να είναι διαθέσιμα αυτά τα χρήματα και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε αρχίσει να αποσύρουμε τα χρήματα από το σύστημα και όχι να χρηματοδοτούμε. Υπάρχει και το θέμα του front loading που σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα χρήματα για το επόμενο τμήμα της χρονικής περίοδος και όπως είπα ήδη μετά το 2014 μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές υπάρχει χρόνος, αλλά μέχρι τότε δεν θα έχουν άμεση επιπτώσεις σε μια κρίση, δεν θα χρειάζονται για την κρίση. Παρ' αυτά, ορισμένε από τι μακροπρόθεσμε επιπτώσει τη κρίση υπάρχουν ακόμα. Απασχόληση Φερρυπίν, η έλλειψη ε, χρηματοδοτικής ε, επένδυσης, κρίση των δημοσίων ε, οικονομικών που διαφέρει από χώρα σε χώρα και έλλειψη διαθεσιμότητας πτώσεων και κεφαλαίου. Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές λοιπόν για μένα είναι συσχετισμός με την Ευρώπη 2020. Θα πρέπει με την χρηματοδότηση αυτή να μην κοιτάμε μόνο την άμεση κρίση, να κοιτάξουμε τις μέσο και μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Δηλαδή μακροπρόθεσμα η φόρο ανάπτυξη και αυτό σημαίνει να εξτάσουμε το δυναμικό ανάπτυξη ε, στα νέα κράτη-μέλη. Οι μακροπρόθεσμες ε, προκλήσεις για τα νέα κράτη-μέλη είναι θέματα ανταγωνιστικότητας και θα πρέπει να δούμε ότι τα μέσα αυτά συνοχής θα πρέπει να είναι ε, τα πιο σημαντικά μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής του 2020. Νέοι ναι, καινοτόμοι μηχανισμοί παραδείγματο χάρη μέσω τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξης, περισσότερο για κεντρικές βασικές πολιτικές, για το μέλλον. Ό,τι θα πανίσουμε από τα μέσα συνοχής θα πρέπει να δούμε ότι θα βελτιώσουμε επίσης τους μηχανισμούς ε, χορήγησης των θεμάτων αυτό, να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση να εξετάζουμε μόνο βραχυπρόθεσμα θέματα, γιατί αυτό δεν είναι καλό και δεν θα είναι η σωστή επιλογή αυτή τη στιγμή. Και δεν θα πρέπει ε, με τα χρήματα αυτά να κλείσουμε κάποια κενά βραχυπράσμα. Θα πρέπει να αρχίσουμε από το μηδέν, να προσανατολίσουμε τα μέσα συνοχής εκ νέου για το 2020 αλλά αυτό μάλλον δεν είναι ε, πολύ σημαντικό γιατί έχουμε το πολυετές ε, οικονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε με τις νέες προοπτικές γιατί χρειάζονται οι πόροι αυτοί, περί τίνος πρόκειται για μετά το 2014, πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε μετά το 2014, ποιος θα είναι ο κύριος τομέας δαπάνης, πώς θα βελ... μεγιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των μέσων αυτών συνοχής και βέβαια τότε θα εξετάσουμε ε, τη συζήτηση για το πόσα χρήματα θα είναι και ποιος θα τα πάρει. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ε, πολιτικές συνοχής λόγω του μεγέθους και της φύσης της να υπάρχουν ισχυρές προότητες, ισχυρή συγκέντρωση Σα είπα τι νομίζω ότι κατά γνώμη μου θα πρέπει να είναι η προτεραιότητε, αλλά αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μα έχει μείνει μισή ώρα για ερωτήσει και απαντήσει. Όποιος θέλει να θέσει ερωτήσει, παρακαλώ να το δηλώσει. Θα κάνουμε δύο γύρους από δύο-τρεις ερωτήσεις στον καθένα. Κύριε Μπέρες. Ευχαριστώ τους δύο εμπειρογνώμονες. Μας διαφώτισαν αρκετά. Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε άλλο τίτλο στο δεύτερο πάνελ. Δηλαδή να πούμε τι μέσα και μηχανισμούς χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη σύγκληση μεταξύ των κρατών Άλλος τίτλος βέβαια επιλέγει. Και η ερώτηση που έχω είναι η εξής. Η κρίση αυτή είτε εντός είτε εκτός της ζώνης ευρώ φωτίζει το, τη βασική πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ο αποκλίνων και όχι ο συγκλίνων χαρακτήρας των οικονομιών. Και όλες αυτές οι στρατηγικές ο στόχο είχαν το να μειώσουν αυτές τις αποκλήσεις και τις διαφορές μεταξύ των οικονομιών. Στις δύο πρόσφατες διευρύσεις υιοθετήσαμε μια στρατηγική που θεωρούσε ότι αρκούσαν τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Αλλά μετά από αυτά που είδαμε και διαπίστωσα ότι ήταν αρκετά συντηρητική η προσέγγιση του κ. Χάιλ, είστε πραγματικά βέβαιος ότι ήταν αρκετά τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Βέβαια, πέραν του σχετισμού δυνάμεων, εσείς ως εμπειρογνώμονας, Θεωρείτε ότι ήταν αρκετά τα κονδύλια του Ταμείου συνοχή. Είναι επαρκή αυτός ο μηχανισμός και γιατί δεν είχαμε καλύτερα αποτελέσματα αν ήταν επαρκή. Στην Ευρωζώνη δεν έχουμε τόσους πολλούς μηχανισμούς σύγκλησης. Έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας, δεν ξέρω αν ήταν αποτελεσματικό. Πάντως, εκτός του, της το Ταμείο Συνοχής ήταν αυτό που θα διευκόλυνε τη σύγκληση. και την ανάκτηση του χαμένου εδάφους από ορισμένε χώρες. Επίσης, ε, έγινε μια διάκριση μεταξύ αλληλεγγύης και ε, μηχανισμών ε, υλοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ο κύριος Ζουλέγκ είπε ότι τα κονδύλια συνοχής προσανατολίζονται περισσότερο στην αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Εγώ περιμένω ότι με την αναθεώρηση αυτή θα προσαρμοστούμε στην συνολική στρατηγική, γιατί τι μας χρειάζονται τα χρήματα αν ε, δεν τα αξιοποιήσουμε για να υλοποιήσουμε τη στρατηγική που αποφασίσαμε και την πολιτική που αποφασίσαμε. Επίσης, ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ποια είναι η γνώμη σας. Και δύο τελευταία σχόλια. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κονδυλίων της συνοχής, πιστεύετε ότι με την κρίση θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια με λιγότερο, ποσο, μικρότερο ποσοστό σε χρηματοδότηση, γιατί αυτή η κατάσταση, η πρόταση κόλλησε στο Συμβούλιο. Πιστεύετε ότι είναι λογική αυτή η θέση του Συμβουλίου με τις νέες χώρες μέλη, άσχετα από το κόστος που θα έχει κάτι τέτοιο για τον προϋπολογισμό των νέων χωρών μελών. Κύριε Ζουλέκ, μάλλον είστε κατά της ε, βραχυπρόθεσμης χρήσης των κονδυλίων της συνοχής. Θεωρείτε δηλαδή ότι τα μέτρα του front loading ε, της προεκταμίευσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ε, ε, εσφαλμένα. κυρία Γιάνσεν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας για το υλικό που μας προσέφεραν, που θα μας βοηθήσει στη συζήτηση και δεν φαντάζομαι να θέλει κανείς να περιορίσει τη χρήση των κονδύλιων συνοχής για τις νέες χώρες μέλη. Εδώ περισσότερο συζητούμε τι θα γίνει στο μέλλον για τις πιο εύπορες και παλιότερες χώρες μέλη. Κύριε Ζούλεκ, είπατε καλύτερα να μείνουμε σε στις βασικές πολιτικές, core policies. Ποιες είναι αυτές οι βασικές πολιτικές, τι πολιτικές εννοείται. Ο κύριος Χάιλ μίλησε ότι χρειάζονται και βασικές πολιτικές, αλλά και ελαστικότητα. Τι αναπρογραμματισμός έγινε, τι ελαστικότητα πιστεύετε ότι χρειάζεται τώρα και τώρα και στο μέλλον. Και εγώ έχω μία σύντομη ερώτηση προς εμπειρογνώμονες. Πιστεύω ότι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι κέριος για τη σύγκληση αλλά και την ανάκαμψη των οικονομιών μας. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις νέες αλλά και για τις παλιές χώρες μέλη. Χρειάζεται για την θέση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την ανάπτυξη και για την ε, τόνωση της κατανάλωσης. Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια συνοχής, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η κυρία Γκέντς. Ευχαριστώ. Θα θέσω την ερώτησή μου στα Ουγγρικά, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Χάιλ, μιλήσατε για τα θεμέλια του Ταμείου Συνοχής. Βέβαια, όταν θεσπίστηκε, όταν ιδρύθηκε το Ταμείο Συνοχής, κανένας δεν περίμενε μια τέτοια κρίση, ούτε φανταζόταν τι επιπτώσεις θα έχει. Τώρα με τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να αντισταθμίσουμε κάπως την κρίση και να βρούμε μηχανισμούς για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της. Επίσης, ανάλογα με την αξιολόγηση που θα γίνει από τη χρήση των μέτρων, θα πρέπει να επαναθεωρήσουμε τη χρήση των ε, μέτρων συνοχής, ιδιαίτερα στο μέλλον αν συνδυάσουμε ή συγκρίνουμε μάλλον τις δύο ομιλίες, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Ο κύριος Χέιλ ισχυρίζεται ότι η πολιτική δυο ομιλιε θα πρέπει να επικεντρωθεί στη σύγκληση, να περιλαμβάνει όλο και περισσότερα κράτη και να αποτελεί το βασικό άξονα και άλλων πολιτικών. Ενώ ο κύριος Ζούλεγκ είπε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σύνεση και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα μέτρα της συνοχής για βραχυπρόθεσμους στόχους. Η στρατηγική του 2020 θα καθορίσει πιο μακρόπνες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. Και θα καθορίσει τη, μελλοντική διαμόρφωση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Πώς πιστεύετε όμως ότι θα πρέπει να μετατοπιστεί η έμφαση της πολιτικής συνοχής. Τι αλλαγές χρειάζονται και πώς θα συνεχιστεί η πολιτική συνοχής υπό το πρίσμα της στρατηγικής του 2020 και πώς εκτιμάται τη στρατηγική του 2020 από αυτή την άποψη. Δεν θέλει άλλος κανεί το λόγο, γι' αυτό και θα δώσω το λόγο στους δύο εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν. Ευχαριστώ. Πολύ εύστοχες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Κυρία Μπέρες, ρωτήσατε αν διαθέτουμε τα απαραίτητα μέσα, τους απαραίτητους μηχανισμούς και αν πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής ε, ανταπεξέλθει στις προσδοκίες που δημιούργησε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. Όταν εξετάζαμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, εννοούσαμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα των κρατικών επενδύσεων στην οικονομία. Η πολιτική συνοχής είναι αποτελεσματική όταν οι πολιτικές που χρηματοδοτούμε με αυτού είναι αποτελεσματικές. Αν γνωρίζουμε πώς θα δημιουργήσουμε πιο βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, πώς θα ενισχύσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και το περιβάλλον, τότε αν οι πολιτικές μας είναι καλές, τότε είναι αποτελεσματική η πολιτική συνοχή. Αν με την πολιτική συνοχή, χρηματοδοτούμε κακές πολιτικές, τότε θα είναι αναποτελεσματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαράζει πολύ αξιόλογες στρατηγικές, όπως τη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά μετά περιμένει από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα μείγμα πολιτικών για να εφαρμόσουν επιτόπου τις στρατηγικές. Από μόνη της η πολιτική συνοχή δεν αρκεί για την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων, ούτε αρκούν τα κρατικά κονδύλια, τα δημόσια κονδύλια για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Φορολογία, υποδομές, πολλές πολιτικές χρειάζονται που εξαρτώνται από τις κυβερνήσεις και από τα εθνικά κοινοβούλια. Η δική τους δράση ε, είναι εξίσου σημαντική όσο και οι πολιτικές συνοχής. Πάντως πιστεύω ότι είναι χρήσιμο αυτό το περίπλοκο εργαλείο της πολιτικής συνοχής και προγραμματίζεται με βάση μακροπρόθεσμη προοπτική και σε, στηρίζεται σε μια οικονομική ανάλυση που μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε μια σαφή γνώμη για το τι θέλουμε να κάνουμε στηρίζεται σε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που είναι χρήσιμη γιατί σημαίνει ότι με την ανάμειξη και των τοπικών φορέων και των περιφερειών έχουμε περισσότερες πληροφορίες από ότι αν στηριχθούμε μόνο στις ε, τομεακές πολιτικές ή στις πληροφορίες που μας δίνουν τα Υπουργεία. Χρειαζόμαστε και την συμβολή των περιφερειών και των τοπικών παραγόντων προγραμματισμός είναι σημαντικό. Η εταιρική σχέση και η μόχλευση που δίνει η πολιτική συνοχή στη χρήση των δημοσίων κονδυλίων, των κρατικών κονδυλίων, αλλά και στα ιδιωτικά κονδύλια, όλα αυτά δημιουργούν ένα μηχανισμό που είναι καλύτερος από οποιοδήποτε άλλο. μέσω του, του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αφιέρωσα πολλά χρόνια στο πρόγραμμα ΦΑΡ, που ήταν ένα πολύ αξιόλογο μέσο. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι ήταν, ε, κατευθυνόταν από ε, τις Βρυξέλλες, κεντρικά, κάτι που το έκανε πιο δίσκαμπτο. Σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη και την ανταγωνιστικότητα και τη σχέση της πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική της Λισαβόνας ή τη στρατηγική του 2020, νομίζω και ελπίζω να ήταν σαφές αυτό που είπα, ότι ήδη από τώρα η πολιτική συνοχή συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική της Λισαβόνας. Όταν σχεδιάστηκαν αυτά τα προγράμματα, υπήρχαν πολλά εργαλεία και πολλοί μηχανισμοί ώστε να μην χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα εφόσον δεν ήταν συμβατό με, τη συνθήκη με την πολιτική της Λισαβόνας. Και αυτή η προσέγγιση στρατηγικού προγραμματισμού του 2007 θα είναι επαρκής και για τα προγράμματα της στρατηγικής του 2020 και δεν υπάρχει καμία αντιδικία μεταξύ του στόχου της σύγκλησης και του στόχου της ε, ε, ανταγωνιστικότητας. Ούτε διαφωνούν τα κράτη-μέλη για την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι οικονομικές πολιτικές και η οικονομική ανάπτυξη. Και υπάρχει συμφωνία προς τους στόχους και της στρατηγικής Λισαβόνας και της στρατηγικής του 2020. Αλλά θα πρέπει ήδη από πριν, σε πολύ πρώιμο στάδιο, να καθορίσουμε με λεπτομέρειες πόσα κονδύλια χρειαζόμαστε για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Έχουμε πόρους, χρειαζόμαστε εμπειρία, χρειαζόμαστε σωστές πολιτικές και ανταλλαγή εμπειριών. Αυτό το κάνουμε στη δική μας ε, κοινότητα. Και πρέπει να αναπτύξουμε και τις εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές, να βελτιώσουμε τις εθνικές αναπτυξιακές πολιτικές. Αναφερθήκατε και στην πρωτοβουλία μείωσης των ποσοστών χρηματοδότηση για του μηχανισμού της ε, πολιτική συνοχή κάτι που κόλλησε στο Συμβούλιο. Όντω ήταν αρκετά τυχή αυτή η συζήτηση. Ήμουν σε μια ομάδα εργασία του Συμβουλίου και δεν υπήρξε καμία συνεννόηση. Μια τέτοια πρόταση που υπευλήθη για να μειωθεί ε, το ποσοστό χρηματοδότηση θα ήταν αρκετά δαπανηρή. υπήρξαν κάποιες προτάσεις από την Ουγγαρία που δεν θα ήταν δαπανηρές από την άποψη, αλλά δεν έγινε σωστή συνεννόηση. Και έτσι μπλοκαρίστηκε αυτό το θέμα. Ελπίζω στο μέλλον να βελτιωθεί η αλληλοκατανόηση. Τώρα, αναπρογραμματισμό και ελαστικότητα. Ερώτηση τη κυρία Γένσεν. Καταρχήν, δεν υπερασπίστηκα την πολιτική συνοχή γιατί φοβόμαι την κατανόμη μεταξύ των νέων χωρών. Ξέρω ότι οποιοδήποτε εμπλεκεί σε μια συζήτηση ε, υπό το πρίσμα των χωρών που είναι συνεισφορείς πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου, όλοι λένε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις νέες χώρες. Αλλά εγώ είπα ότι έχουμε στα χέρια μας μια πολιτική που δεν ε, πρέπει να περιοριστεί στην αλληλεγγύη. Θα, είναι, θα χρησιμοποιηθεί και ως μηχανισμός αλληλεγγύης, αλλά δεν εξαντλείται εκεί ο ρόλος του. Και είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι η επανεθνικοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής και η συμπερίληψη των χωρών μπορεί να τη, χρηματοδο... χρηματοδοτήσουν, γιατί πολύ συχνά αναφέρεται γιατί να στέλνουμε χρήματα στις Βρυξέλλες και μετά να τα παίρνουμε πίσω αφού περάσουμε από όλα τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ενώ θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Λάθος. Κοιτάξτε την Ιρλανδία. Από το 2000 έως το 2006 είχαν εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα αξία 56 δισεκατομμύριων ευρώ. Ξέρετε πόσα ήταν κοινοτικά κονδύλια. 8 δισεκατομμύρια, ένα μικρό τμήμα δηλαδή. Για όλες τις χώρες, είτε αυτές που συνεισφέρουν ή αυτές που είναι δικαιούχοι αποδέκτες, υπάρχει δυνατότητα να αποτελέσει η στρατηγική του 2020 βάση για τις εγχώριες πολιτικές, ακόμη και για εκείνες που χρηματοδοτούνται εθνικώς. Η στρατηγική του 2020 και οποιαδήποτε κατευθυντήρια γραμμή θα προκύψει από την πολιτική συνοχή δεν ε, χρειάζεται να περιοριστεί στα κοινοτικά κονδύλια. Αν συνδυάσουμε τις εθνικές με τις κοινοτικές προσπάθειες, τότε θα έχουμε καλύτερες αναπτυξιακές πολιτικές που θα υλοποιούν τους κοινοτικούς στόχους. Και αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, χρειάζεται σωστή αξιοποίηση των πόρων μας, αρκεί να διδαχθούμε τα παθήματα, από τα παθήματα της κρίσης και από τα επιτέγματά μας από το 2007. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι πολύ σημαντικέ ήταν οι πρωτοβουλίε του Τζέρεμι το 2007. Δεν ήταν εύκολο να αναγνωριστεί ακόμη και στην Ουγγαρία ότι χρησιμοποιούνται καλύτερα, ότι βοηθούνται καλύτερα από ε, επιδοτήσεις που επιστρέφονται και όχι μόνο από δωρεάν επιδοτήσεις και χρειάζονται προϋποθέσεις θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναλάβουν τις δεσμεύσεις της διεύρυνσης τους, της εξάπλωση των δραστηριοτήτων τους και της διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Με τις πολιτικές συνοχής ε, έχουμε πολλούς μηχανισμούς εγγυήσεων και παροχής δανείων, Πάντως ε, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση του μηχανισμού Τζέρεμι και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας άνοιξε τα μάτια για την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, υπάρχει αντίφαση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων σύγκλησης και συνοχής. Θα ήθελα να σας πω, κυρία Γκέντς, κύριε Υπουργέ, ότι και εγώ και ο κύριος Ζουλέκ είπαμε ότι η πολιτική συνοχή μπορεί να είναι το σημαντικότερο εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε και οι δύο και αυτό ήταν το πιο σημαντικό από τι ε, ομιλίε μα. Κύριε Ζουλέκ, θέλετε να προσθέσετε και στα σχόλιά σα. Σχετικά με το αν διαθέτουμε του μηχανισμού για να βελτιώσουμε τη συνοχή έχουμε αρχή των μηχανισμών αυτών, αλλά δεν είναι επαρκής για την ώρα. Το γενικό πρόβλημα που έχουμε στο επίπεδο της Ένωσης είναι ότι συχνά βάζουμε υπερβολικά φιλόδοξους στόχους και μετά δεν θεσπίζουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Επανέρχομαι σε αυτό που είπε για την Ευρώπη 2020. Αυτή είναι και η βασικότερη πρόκλησή μας για το 2020. Όχι μοναχά να αποφασίσουμε το ποιοι θα είναι οι στόχοι, αλλά να καταστήσουμε σαφές τι θα χρειαστεί για να επιτύχουμε τους ε, ε, στόχους αυτούς Ποια είναι διαθέσιμα. Η πολιτική συνοχή είναι ένα από τα μέρη αυτά, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί. Υπάρχει, υπάρχουν ορισμένε ε, ορισμένοι τομεί όπου ακόμη δεν διαθέτουμε του απαραίτητου μηχανισμού. Ένα που νομίζω ότι είναι σημαντικό στη συζήτηση περί συνοχή, περί συγκλήσεω περισσότερο για νέε χώρε μέλη, όπου είναι πολύ χαμηλές ακόμα οι επενδύσεις σε θέματα παιδείας, κατάρτισης και αγοράς εργασίας. Το κοινωνικό ταμείο από μόνο του δεν αρκεί, θεωρώ εγώ, για να ε, μπορέσει σε αυτό να βασιστεί η αλλαγή που είναι απαραίτητη για το μέλλον. Για το μέλλον αυτό που ε, χρειάζεται είναι να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και για τις παλιές αλλά και για τις νέες χώρες μέλη. Νομίζω ότι αφενός χρειάζεται σύγκληση Αφενός χρειάζεται προσπάθεια βελτίωση του βιωτικού επέδου σε όλες τις χώρες μέλη αν θέλουμε να αυξήσουμε εν τέλει το ρυθμό ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, είναι κρίμα που δεν επετεύθη συμφωνία. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Όμως όταν αντιμετωπίζουμε κρίση όπως η παρούσα, πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε με πιο εύκαμπτο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία που διαθέτουμε. Και αυτό ισχύει και για τα ταμεία τα οποία, τα κονδύλια που δεν έχουν ακόμα δαπανηθεί και που υπάρχουν στον προπολογισμό. Και αυτά πρέπει να διατεθούν με σωστό τρόπο. Σε αυτούς τους τομείς μπορούμε νομίζω να βελτιώσουμε την απόδοσή μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα το front loading ήταν σφάλμα. Εγώ δεν είπα πολύ ξεκάθαρα άποψη. Δεν θεωρώ ότι το front loading ήταν την εποχή που θεσπίστηκε λάθος. Νομίζω πάντως ότι τώρα πλέον δεν είναι ορθό. Γιατί έχουμε τώρα τις αποσύρσεις των ε, χρημάτων που δόθηκαν για κίνητρα και πρέπει να δούμε αν η κρίση θα αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. Αν είναι βραχυπρόθεσμη, τότε είναι πραγματικά σωστό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γεφυρώσουμε αυτό το βραχυπρόθεσμο διάστημα. Αν μιλούμε για μακροπρόθεσμη ωστόσο κρίση, τότε δεν αρκεί, διότι θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα μακροπροθεσμότερα, χωρί όμω διαθέσιμα τα ίδια κονδύλια για να κάνουμε front loading. Οι λεγόμενε co co-policies, αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένω ήταν ότι αυτά που βλέπουμε περισσότερο είναι οι πολιτικές χρηματοδότησης των χωρών μελών που θα ήταν πιο προσαρμοσμένες στις καθημερινές τους πολιτικές. Δεν είναι νέες πολιτικές, είναι πάντως αυτά που αναμένει το κοινό να πράξει μια χώρα, ένα κράτος για και μεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό το, το θέμα που τίθεται είναι των οργανισμών που ε, διαθέτουν εν τέλει τα κονδύλια για τις χρηματοδοτήσεις, ποιος δηλαδή δίνει τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα και πόσο κοντά είναι στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε νέα, νέους μηχανισμούς με χορήγηση δανείων και νομίζω επίσης ότι και οι έμεσε επενδύσει για την βελτίωση δηλαδή των προσόντων των ε, εργαζόμενων ή αυτών που επιθυμούν να βρουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, πρέπει να αυξηθούν. Αυτή τη διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμου και προκοπρόθεσμου δεν τη θεωρώ αντίφαση. Αν θέλουμε να εξετάσουμε το πιο μακροπρόθεσμο μέλλον που θα, βρούμε, που θα δούμε την σύγκριση, που θα δούμε την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των χωρών μελών. Αφενός χρειάζεται να εγκύψουμε στα βραχυπρόθεσμα προβλήματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση, αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να επενδύσουμε σε πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν σε οικονομική αύξηση. Και αυτό με ορίζοντα την Ευρώπη του 2020 και φροντίζοντας ώστε να έχουμε αυτή τη φορά μια ε, στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης η οποία να μπορέσει να ε, επιτρέψει την επίτευξη των στόχων που έχουμε θεσπίσει. Η κυρία Χιούπνερ έχει μια τελευταία ερώτηση. Έχει το λόγο κυρία μου. Μια ερώτηση αν με επιτρέπετε ακόμα γιατί υπάρχει λίγος χρόνος. Μπερδεύτηκα λίγο όταν μιλήσατε για front loading σαν stimulus package, σαν ε, ε, δέσμη μέτρων ε, κινήτρων. Ήταν ένα από τα πρόσθετα ωφέλη που δόθηκαν στις χώρες μέλη μέσα στα υφιστάμενα προγράμματα ωστόσο και ήταν αφιερωμένο στην εφαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων. Δεν δημιούργησε νέα μέτρα επενδύσεων, νέες παρεμβάσεις σε επενδύσεις εντελώς έξω από αυτά. Ε, με εξέπληξε το σχολείο σας και ίσως μπορείτε να το διευκρινίσετε. Δεύτερο, μια ερώτηση προς εσάς. Υπάρχουν πολλές αδυναμίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ίσως να μην είναι τώρα ο τόπος και ο χρόνος για να τα συζητήσουμε. Πάντως, ένα από τα στοιχεία που διαπιστώνω είναι ότι η στρατηγική αυτή δεν λαμβάνει διόλου υπόψη της την ανομοιομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιφερειακή σκοπιά λοιπόν είναι παράξενο το έγγραφο αυτό, διότι δεν κάνει διαφοροποίηση της Ευρώπης, ε, ε, οικονομικά μιλώ, από την ε, σκοπιά του δυναμικού ανάπτυξης, αλλά και των προβλημάτων ανάπτυξης. Διαρωτώμε, δε, εάν αυτή η στρατηγική η οποία δεν επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι, τη διαφοροποίηση δηλαδή, την διαφορετικότητα της Ευρώπης, μήπως είναι τυφλή απέναντι στις περιφερειακές διαφορές. Έρχομαι και πάλι σε αυτό το σύνδεσμο μεταξύ της Ευρώπης 2020 και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Όταν θέτω το ερώτημα γιατί η πολιτική συνοχής ήταν τόσο σημαντική για την ανάκαμψη τον Νοέμβριο του 2008, λόγω της ικανότητάς της δηλαδή, όπως είπατε και οι δυο σας, να συνδεθεί το βραχυπρόθεσμο πακέτο με τους ε, μακροπρόθεσμους στόχους της ανάπτυξης και της ε, μεταλλαγής αυτής. Ε, ήταν βασισμένο σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική ανάπτυξης και οι χώρες μέλη ήταν, είχαν αναλάβει, είχαν δεσμευτεί να βρουν την χρηματοδότηση. Τώρα αυτή η διασύνδεση με, την, τον ορίζοντα 2020 μου φαίνεται φυσική και σημαντική για την Ευρώπη. Λόγω των συνδέσμων που μπορεί να προσφέρει η πολιτική αυτή. Και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για τους μηχανισμούς επίτευξης των στόχων που πάλι λείπουν από τη στρατηγική του 2020. Εάν συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την τομεακή αυτή προσέγγιση, διότι αυτό προτείνει η Ευρώπη του 2020, είναι στην πραγματικότητα τομεακή προσέγγιση στην ε, ανάπτυξη, η οποία μετά θα μεταφραστεί και σε τομεακού προπολογισμού τη Ευρώπη κάτι που θα μας οδηγήσει σε 20 χρόνια πίσω το λιγότερο. Ή θα σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε 100% earmarking για κάθε νέο μηχανισμό που θα δημιουργείται αφού ο κάθε μηχανισμός αυτός θα είναι αφιερωμένο σε συγκεκριμένα πράγματα. Ή υπάρχει αρχικη επιλογή, οι πολιτικοί μηχανισμοί, ε, η πολιτική μάλλον, να δώσει τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να διαθέτουν μια ευκαμψία που νομίζω ότι θα είναι απαραίτητη, διότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Και μάλλον χρειαζόμαστε διαφορετική παλέτα παρεμβάσεων. Σε κάθε μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, να σας παρακαλέσω να κάνετε σχόλια. Αν θα πρέπει να επιλέξουμε την τομεακή αυτή προσέγγιση με 100% earmarking ή μια πολιτική συνοχής με κάποια περιθώρια ελιγμών, κάποια περιθώρια ε, ελιγμών παρέμβασης. Πολύ σημαντικά ερωτήματα, κυρία Χιούπνερ μου, αλλά φοβούμαι ότι ε, μέσα σε 1,5 λεπτό που έχουν οι ε, εμπειρογνώμονες δεν θα προλάβουν ίσως να τα απαντήσουν όλα. Ναι, ναι. Θα ήταν μέγα ασφάλμα να υιοθετήσει κανείς μια ε, στρατηγική που να είναι τυφλή απέναντι στις περιφερειακές διαφορές. Θα έπρεπε να υπάρξει ένας μηχανισμός θα ήταν λάθος μάλλον. Θα ήταν λάθος να υπάρξει μια τομιακή προσέγγιση χωρίς να εξετάσει το τι συμβαίνει επί τόπου. Για παράδειγμα, πράσινη οικονομία. Ποιος θα είναι ικανό στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ε, να θεσπίσει το μηχανισμό που ορισμένοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει για τις περιβαλλοντικές επενδύσεις ε, στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο αυτοί που είναι επιτόπου. Έκανα μερικά ταξίδια στην Αυστρία, στην ε, ε, περιοχή που λέγεται Στάιρ και κάθε μια από τις κοινότητες, αυτό αποκαλείται εκεί κοινότητα κλίματος. Κάνουν δηλαδή πράγματα επιτόπου για να προωθήσουν πράγματα που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Καλύτερο αυτό παρά μια ε, σούπερ πολιτική που να ε, επιβάλλεται άνωθεν από τις Βρυξέλλες. Και σε ό,τι αφορά την ευκαμψία ή ευελιξία, flexibility, νομίζω ότι υπάρχει μια θεμητή ανησυχία ότι δεν μπορεί κανείς ε, να δώσει από πολύ λίγα σε πάρα πολλούς. Οι προτεραιότητες των χωρών θα είναι συνήθως αυτές που περιλαμβάνονται στη στρατηγική του 2020. Αλλά πώς θα εφαρμοστούν. Αυτό πρέπει να κριθεί επιτόπου από κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Πάλι αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει η πολιτική συνοχή, όμως, όχι όμως οι τομεακές πολιτικές. Ζούλεγκ. Για το front loading, αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω πριν είναι ότι το front loading δόθηκε για να διατηρηθεί μια οικονομική δραστηριότητα επειδή υπήρχε έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας ή ιδιωτικής σύντησης, εάν θεωρούμε ότι είναι βραχυπρόθεσμη η κρίση και αυτή η ιδιωτική δραστηριότητα θα ανακάμψει τα επόμενα χρόνια, τότε έχει νόημα να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο front-loading, γιατί αργότερα τότε μπορούμε, όταν θα αρχίσει να δραστηριοποιείται ξανά η ιδιωτική δραστηριότητα, δεν θα υπάρχει πια, δεν θα είναι τουλάχιστον αισθητή η έλλειψη ε, κονδυλίων, γιατί θα έχει ε, ε, δραστηριοποιηθεί ο ιδιωτικό τομέας. Αν μιλάμε όμως για διαρκέστερη μείωση τη οικονομικής δραστηριότητα, τότε δεν έχει νόημα να δώσουμε τόσο πολύ έμφαση στο front loading γιατί θα αντιμετωπίσουμε πολύ βαρύτερα προβλήματα όταν θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα μας τελειώσουν τα λεφτά. Για την Ευρώπη 2020 συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να δώσουμε στις χώρες μέλη και στις περιφέρειες την ευκαμψία να μπορούν να αποφασίζουν πού θα ρίξουν την έμφαση. Αυτό χρειάζεται, που χρειάζεται είναι μια συμφωνία στους γενικούς στόχους και ελπίζω να προκύψει από την Ευρώπη 2027, αλλά βέβαια ε, ακόμα έχει πολλές ελλείψεις το υφιστάμενο σχέδιο και ελπίζω ότι θα περάσει από διάφορες αναθεωρήσεις με τις οποίες θα το φτάσουμε στη τελική του μορφή, αλλά αυτό θα είναι το βασικό εργαλείο που θα ριξουν την εμφαση αυτο χρειαζεται που χρειαζεται ειναι μια συμφωνια στους γενικους στοχους και ελπιζω να προκυψει απο την ευρωπη 2027 αλλα βεβαια ακομα εχει πολλες ελλειψεις το υφισταμενο σχεδιο και ελπιζω οτι θα περασει απο διαφορες αναθεωρησεις με τις οποιες θα φτασουμε στη τελικη του μορφη αλλα αυτο θα ειναι το βασικο εργαλειο που θα χρησιμοποιηθει και τώρα περιφέρειες και χώρες μέλη. Ναι, θα πρέπει να είναι και υπόλογα για την επίτευξη των στόχων και να δείξουν ποιους μηχανισμούς θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα για να επιτύχουν τους στόχους που έχουν καθορίσει. Και νομίζω ότι αυτό δεν το έχουμε για την ώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Ζούλε και ευχαριστώ όλες και όλους τους αγορητάς, ευχαριστώ και όλες και όλους τους συναδέλφους. Νομίζω ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποδοτική η συζήτηση. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, διερμηνείς ευχαριστούν την Πρόεδρο. Το τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεως είναι η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίας που θα είναι η 11η Μαρτίου στο Στρασβούργο, όπου θα συζητήσουμε το θεματικό κείμενο για την, τα μελλοντικά μοντέλα της Financial Supervision και μετά στις 18 Μαρτίου στις Βρυξέλλες όπου θα κάνουμε την πέμπτη δημοσία κρόαση για την ε, ε, European Economic Governance και για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. Σας ευχαριστώ.